Λοιπόν, ξεκινάμε τη συνεδρίαση. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλωσορίζουμε θερμά στη σημερινή συνεδρίαση. Έχουμε λοιπόν το σχέδιο της ε, ημερήσιας ε, διάταξης, ε, το οποίο σας διανεμήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου και Όσον αφορά την ημερησία διάταξη, θα έχουμε και ένα νέο σημείο, το 45, που είναι το πρόγραμμα εργασίας και την ενδιάμεση ανασκόπηση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ε, αυτό θα το εξετάσουμε αμέσως μετά το σημείο 42, λέει ο Πρόεδρος. Συμφωνείτε πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο σημείο, που πρόκειται για την... Ε, έγκριση των πρακτικών της 19ης και 20 Ιανουαρίου του 2009 τα οποία πρακτικά διανεμήθηκαν στις 6 ε, Φεβρουαρίου. Τώρα θα ήθελα να ζητήσω τη συνένεσή σας ε, για ένα θέμα, αγαπητοί συνάδελφοι, για το εξής δηλαδή. Πρόκειται για συζητήσεις ε, που έχουν σχέση με την Επιτροπή των Περιφερειών και με τον ε, αστυνομικό οργανισμό. Οι συζητήσεις αυτές ε, θα συνεχίζονται μέχρι αύριο το μεσημέρι. Δηλαδή, ο αρμόδιος εισηγητής, ο κύριος, οι κύριοι Σίντεγκαρτ και Φέλνερ, ακόμα διεξάγουν τις διαπραγματεύσεις. Ενδέχεται λοιπόν αυτό τα δύο σημεία της ημερήσιας ε, διάταξης ε, να πρέπει να συζητηθούν και κλεισμένων των θυρών. Συμφωνείτε εσείς επ' αυτού. Ε, στην περίπτωση βέβαια, όπως σας είπα, κατά την οποία οι συγητές ζητήσουν και οι ίδιοι να συζητηθεί το θέμα και κλεισμένων των θερών. Υπάρχει κάποιος που να διαφωνεί, από ό,τι βλέπω όχι. Σας ε, ευχαριστώ πολύ για τη διευκόλυνση της ε, διαδικασίας. Σας είπα πρόκειται για αυτούς τους δύο οργανισμούς. Πάμε στο σημείο υπαριθμών 3 της ε, ημερήσιας διάταξης. Οι γλώσσες διερμηνίες υπάρχουν στο ενημερωτικό δελτίο και θα ήθελα να σας ανακοινώσω το κύριε Κυρίτα και Ντέιβιτ αναπληρωματικά μέλη θα γίνουν αναπληρωματικά μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και ο κύριος Σουλόνς ε, θα γίνει ε, αναπληρωματικό μέλος ε, της Επιτροπής μας εκ μέρους της Σοσιαλιστικής Ομάδας. Θα ήθελα επίσης να σας ανακοινώσω ότι αυτή η συνεδρίαση όπως συνέβη και με την προηγούμενη θα μεταδίδεται μέσω του web stream σε ολόκληρο τον κόσμο αυτό, όσον αφορά το θέμα αυτό, μπορείτε στο σημείο υπαριθμών 3 να βρείτε όλες τις σχετικές λεπτομέρειες. Θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή σε μια ομάδα εργασίας που αποφασίσαμε στις 4 Νοεμβρίου. Εκεί θέλουμε να ασχοληθούμε με τα διοικητικά στα ίδια τα κράτη-μέλη και ε, τούτο ως follow-up των ε, ερευνών της Όλαφ. Ξέρετε ότι αρμόδιο μέλος είναι η κυρία Γκρέσλα στις 19 Φεβρουαρίου στην αίθουσα ISB 1G2 από τις 2 ε, μέχρι τις 5.30 θα συνεδριάσει η ομάδα και βέβαια είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Έχετε κάτι να πείτε για την ημερησία διάταξη από ό,τι βλέπω. Όχι, πάμε λοιπόν στο σημείο υπαριθμών 4 της ημερησίας διάταξης που είναι πολύ σημαντικό. Πρόκειται για την απαλλαγή του ή απαλλαγές του 2007, παρουσίαση της ε, σύστασης του ε, Συμβουλίου και εδώ θα ήθελα να καλωσορίσω τον Προεδρεύοντα, τον κύριο Μύροσλαβ Κάλουσεκ από τη Δημοκρατία της Τσεχίας. Ε, σας καλωσορίζουμε θερμά κύριε Υπουργέ και έχετε ευθύς αμέσως το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ναι, Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητέ κύριε Κάλλας, Αγαπητοί βουλευτές, θέλω να σας πω ότι για μένα είναι μεγάλη τιμή και χαρά το γεγονός ότι έχω τη δυνατότητα σήμερα εκ μέρους του Συμβουλίου να σας παρουσιάσω τη σύσταση της Κομισιόν για τις απαλλαγές του 2007. Αυτή η σύσταση πέρασε από το ΕΚΟΦΗΝ στις 10 Φεβρουαρίου και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι αυτό το βρίσκω ιδιαίτερα θετικό. Το Συμβούλιο βρίσκει σημαντικό το γεγονός ότι το ελεγκτικό συνέδριο τοποθετήθηκε θετικά όσον αφορά το κλείσιμο των ισολογισμών. Και θέλω να σας πω ότι αυτό συνέβη χωρίς κανενός είδους επιφύλαξη. Το Συμβούλιο λοιπόν καλεί την ε, Κομισιόν να συνεχίσει να εγγυάται την υψηλή ποιότητα των λογιστικών. Θεωρώ λοιπόν ότι εδώ είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η ε, Κομισιόν εισήγαγε το σύστημα του accrual accounting μόλις το 2005. Και βλέπουμε λοιπόν ότι το σύστημα αυτό λειτουργεί πολύ καλά. Το Συμβούλιο διαπιστώνει ότι ε, το ελεγκτικό συνέδριο δεν έχει καμία επιφύλαξη όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες. Παράλληλα, το ελεγκτικό συνέδριο διαπιστώνει ότι λειτουργήσαν σωστά τα συστήματα ελέγχου. Θετική είναι και η τοποθέτηση όσον αφορά τα λογιστικά. Βλέπουμε ότι ο κανισμός 1-2 βοήθησε στο να διεκπαιρώνονται ταχύτερα οι υποχρεώσεις. Παρόλα αυτά, ε, παρά αυτές τις ε, θετικές διαπιστώσεις του Συμβουλίου. Εκείνο που είναι λυπηρό είναι ότι οι περισσότερες ε, δαπάνες επηρεάζονται αρνητικά και θα ήθελα να σας ε, αναφέρω την ε, διαπίστωση του Συμβουλίου όπου εκφράζει ε, την ε, λύπη του για το ότι όσον αφορά τη δήλωση της αξιοπιστίας υπάρχουν επιφυλάξεις σχετικά με το 2007 και παρά τα μέτρα που ελήφθησαν έτσι ώστε να βελτιωθούν τα συστήματα ελέγχου. Το ελεγκτικό λοιπόν συνέδριο καλείται να ε, το Συμβουλίο να τοποθετηθεί γενικότερα για άλλη μια φορά στο θέμα της ε, γεωργίας, της ε, ενέργειας, των μεταφορών, των εξωτερικών σχέσεων. Σε αυτούς τους τομείς το ελεγκτικό συνέδριο δήλωσε ότι τα συστήματα ελέγχου και εποπτείας δεν είναι απόλυτα παρά μόνο εν μέρει αποτελεσματικά. Το Συμβούλιο διαπιστώνει ότι οι περισσότερες δαπάνες ε, ε, εκταμιεύθηκαν από το ε, Ταμείο Εγγύησεων το 2007 και με λύπη του το Συμβούλιο διαπιστώνει ότι όσον αφορά τις πληρωμές τα περισσότερα λάθη εντοπίζονται στη γεωργική ανάπτυξη και υποθέτουμε ότι τούτο οφείλεται στο ότι οι κανόνες είναι ιδιαίτερα περίπλοκοι. Όσον αφορά τώρα τις δαπάνες στον τομέα της ε, συνοχής, το Συμβούλιο ε, διαπιστώνει ότι ε, γίνεται λόγος για τις δαπάνες μόνο για τη χρονική περίοδο 2000 έως 2006. Εκεί έλαβαν χώρα περισσότερες δαπάνες και το Συμβούλιο ανησυχεί για την ε, δήλωση του ελεγκτικού ε, συνεδρίου. Στις δαπάνες εντοπίζονται αρκετά λάθη και τα συστήματα ελέγχου και εποπτείες είναι μόνο εν μέρη αποτελεσματικά. Εξάλλου το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνεχής, συνοχής είναι ε, πολυετής. Ε, οι έλεγχοι ε, συνεχίζονται, δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Θα έλεγα λοιπόν, εγώ θα πρότεινα το ποσοστό των λαθών να το λάβουμε υπόψη μας γιατί δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Και θα ήθελα να κάνω και μια παρατήρηση που είναι πολύ σημαντική για το Συμβούλιο. Δηλαδή, στο πλαίσιο της βελτίωσης βελτίωσης ε, της ε, δημοσιονομικής ε, διαχείρισης και των ευθυνών για κοινή διαχείριση διαπιστώνουμε ότι πράγματι οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι εργάστηκαν αποτελεσματικά, συνεργάστηκαν σε όλα τα επίπεδα ελέγχου και διαχείρισης. Και εδώ το Συμβούλιο υπενθυμίζει το ρόλο κλειδί των κρατών μελών όσον αφορά τη βελτίωση της ε, δημοσιονομικής ε, διαχείρισης. Επίσης ε, υπενθυμίζει τα εσωτερικά συστήματα ελέγχου. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω και τους ε, ετήσιους ελέγχους των κρατών μελών. Ε, το Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ελέγξει την συμβατότητά τους ε, με τις διοργανικές συμφωνίες και με το δημοσιονομικό κανονισμό. Θα ήθελα τώρα να επιστήσω την προσοχή σας σε ορισμένες προτεραιότητες του Συμβουλίου με στόχο να ελέγξουμε το κόστος σε σχέση με την εποπτεία και τον έλεγχο. Έχοντας κατά νου ότι οι επιπτώσεις ε, μετά από τον εντοπισμό λαθών καθίσανται σαφείς μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Το Συμβούλιο λοιπόν ε, προτείνει να καθοριστούν συγκεκριμένες διαδικασίες και αυτές να ακολουθηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων. Όσον αφορά τη συνοχή, το Συμβούλιο ε, χαιρετίζει τα μέτρα τα οποία λήφθησαν στο πλαίσιο του ε, οικονομικού προγράμματος που έχουμε καθορίσει. Εδώ συμπεριλαμβάνονται και τα εφάπαξ ε, ποσά. Ε, το Συμβούλιο καλεί την Κομισιόν ε, σε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη να συνεχίσει τις προσπάθειές της και να αναζητήσει περαιτέρω δυνατότητες απλούστευσης. Πριν λοιπόν τελειώσω με την παρέμβασή μου, θα ήθελα να συστήσω την απαλλαγή για ε, εκείνους τους οργανισμούς που έχουν μία νομική οντότητα και που ε, χρηματοδοτούνται από τα κράτη-μέλη. Παρότι στον ε, τομέα της ε, οικονομικής διαχείρισης ε, των εκτελεστικών οργανισμών υπάρχει κάποιο περιθώριο χειρισμών. Πάντως ε, το Συμβούλιο συστήνει να χορηγηθεί η επαλλαγή σε όλους αυτούς τους οργανισμούς. Επίσης το Συμβούλιο συστήνει την απαλλαγή τριών άλλων εκτελεστικών οργανισμών με βάση τη δήλωση αξιοπιστίας του ελεγκτικού συνεδρίου. Και θα ήθελα ε, τελειώνοντας να σας πω ότι η, ε, ο, ο έλεγχος, η, αναθεώρηση του 2007 έγινε έχοντας ε, κατά νου τις προσπάθειες που καταβάλλονται έτσι ώστε να γίνεται σωστή χρήση των κοινοτικών κονδυλίων. Το Συμβούλιο λοιπόν είναι σε θέση να προτείνει την γενική απαλλαγή για τον Προεπλογισμό του 2007. Αυτή είναι η σύσταση του Συμβουλίου. Και εγώ βεβαίως βρίσκομαι εδώ μπροστά στο Κοινοβούλιο. Η απόφαση του Κοινοβουλίου είναι κυρίαρχη απόφαση. Εσείς τελικά είστε εκείνοι που θα πείτε τον τελευταίο λόγο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την παρουσίαση και θα έλεγα ως συνήθως... Ε, Πρώτα απ' όλα να δώσουμε το λόγο στους ε, επίσημους εισηγητές μας το 2007 και μετά να ξεκινήσει η συζήτηση. Κύριε εισηγητά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα κύριε Υπουργέ για την παρουσία αυτή που μας κάνετε εκ μέρους του Συμβουλίου. Θέλω να σας πω και εκ μέρου εμένα προσωπικά αλλά και των συναδέλφων ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε εδώ όταν συζητάμε για την απαλλαγή όταν πρόκειται για ολόκληρο το Κοινοβούλιο γιατί είναι πολύ καλό να υπάρχει διάλογο, συζήτηση μεταξύ των δύο βραχιών έγκριση του προπολογισμού και της Κομισιόν. Τώρα, από αυτά που είπατε, αναφερθήκατε στο ποσοστό του 11%, ποσοστό λάθους για τη συνοχή που πρέπει με κάποια επιφύλαξη να το δούμε. Σύμφωνα με το κείμενο του ελεγκτικού συνεδρίου δεν πρόκειται για ποσοστό σφάλμα, αλλά πρόκειται για τα ποσά τα οποία κακώς επεστράφηκαν. Είναι τελικά ποσοστό σφάλματος ή είναι ε, κατά λάθο επιστροφές. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα και θέλουμε να ξέρουμε περί τίνο πρόκειται. Επίσης θέλουν να μας πείτε για τις εθνικές δηλώσεις αξιοπιστία των κρατών μελών. Γιατί όσο περνά ο καιρό, εμείς τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι τα κράτη-μέλη διστάζουν, αρνούνται, ορισμένα τουλάχιστον. Εσείς πώς βλέπετε το μέλλον των εθνικών δηλώσεων. Το Κοινοβούλιο θέλει να υπάρχουν διότι αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα με, την, τον επιμερισμένο έλεγχο. Εμείς δεν εκπροσωπούμε τη μία την άλλη χώρα. Το Συμβούλιο όμως ενδιαφέρεται περισσότερο για αυτό το θέμα των εθνικών δηλώσεων. Λοιπόν, θέλω να ξέρω τη γνώμη σας επίσης για την ποιότητα των ε, εκθέσεων ελέγχου που γίνονται κάθε χρόνο και που σας στέλνουν οι εθνικές δηλαδή δικήσεις. Ξέρω ότι η ποιότητα διαφέρει και πολλές φορές δεν είναι στο ύψος που θα έπρεπε. Τρίτο θέμα. Για το ανεκτό ε, ποσοστό σφάλματος. Το ελεγκτικό συνέδριο μας έχει στείλει πολλά και διαφορετικά μηνύματα από αυτού. Η Κομισιόν μας έστειλε μια ανακοίνωση η οποία επί της ουσίας θεωρεί ότι οι πολιτικοί θα αποφασίσουν το ανεκτό ποσοστό σφάλματος. Ποια είναι η δικιά σας η άποψη από αυτού. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι πολύ επικίνδυνο να είναι οι πολιτικοί οι οποίοι θα ανακατευτούν στη μεθοδολογία ελέγχου. ελέγχου. Γιατί η εκτίμηση του ποσοστού λάθους έχει να κάνει με την ίδια τη μεθοδολογία του ελέγχου. Τέλος, Θέλω την άποψή σας, κύριε Υπουργέ, για κάτι που έχει να κάνει με αυτό στο οποίο θα έρθω σε λίγο, αλλά υποφελούμε από την παρουσία σας εδώ, μια που ξέρω ότι σε λίγο θα φύγετε, για να μου πείτε το εξής. Τι λέτε εσείς για να βάζαμε περισσότερο τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια να ανακατευτούν στη διαδικασία απαλλαγής. Αυτό βέβαια τι σημαίνει. Σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να συμφωνήσουν, καταρχήν, ώστε να είναι τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια τα οποία να μπορούν να δίνουν ε, δηλώσεις ελέγχου που να τηρούν βέβαια τις προδιαγραφές που πρέπει. Τα κράτη-μέλη δεν είναι δυνατόν να λένε συγχρόνω δεν θέλω να υπογράφω εθνικέ δηλώσει αξιοπιστία και συγχρόνω να μην βάζουν εθνικά όργανα ελέγχου ανεξάρτητα, όπω είναι τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια, να δουλεύουν προ αυτή την κατεύθυνση. Δεν γίνεται. Για όλα αυτά θέλω τη γνώμη σα και σα ευχαριστώ για άλλη μια φορά που ήρθατε. κύριε Πρόεδρε, αν θέλετε μπορείτε να απαντήσετε. Καταρχήν ε, ευχαριστώ για τις ε, ερωτήσεις που μου κάνατε και <clears throat> φαντάζομαι θα μου επιτρέψετε να σας πω το εξής. Πολλές φορές ε, με κάλεσαν να πω και εγώ τι σκέπτομαι. Συγκεκριμένα όταν ανέλαβα τη θέση του προεδρεύοντος του ΕΚΟΦΗΝ εγώ είχα υποσχεθεί ότι την προσωπική μου άποψη θα την απέκρυπτα και θα προσπαθώ στο βαθμό του δυνατού να αναφέρω την θέση του Εκοφήν, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου. Ε, δεν πρέπει να εκφράζω προσωπικές και εθνικές απόψεις, αλλά να συντονίζω τις απόψεις του ΕΚΟΦΗΝ με στόχο να επιτύχω τη συνένεση. Αυτή είναι η υποχρέωσή μου. Κατά τα ε, και για αυτό το λόγο μάλλον σας λέω ότι είμαι υποχρεωμένο να υπερασπιστώ τη θέση του Συμβουλίου. Όσον αφορά την ε, πρώτη ερώτηση που μου κάνετε σχετικά με το ποσοστό ε, λαθών ε, της τάξης του 11% και κατόπιν θα πρέπει να εκταμιεύονται τα κονδύλια ή όχι. Εδώ θέλω να πω ότι το ελεγκτικό συνέδριο δεν είναι υποχρεωμένο να λάβει, να λάβει απόφαση για ένα συγκεκριμένο έτος. Ισχύει δηλαδή το εξή ε, στη συγκεκριμένη περίπτωση ισχύει, ισχύει το ποσοστό του 11% λαθών, άρα δηλαδή δεν θα έπρεπε να χορηγηθούν το 11% των ε, κονδυλίων. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να έχετε πάντα κατά νου ότι πρόκειται για πολιετή προγράμματα τα οποία θα συνεχιστούν και πάρα πολλά λάθη είναι δυνατόν να διορθωθούν. Τώρα, ε, ποιο ήταν ε, πραγματικά το ποσοστό του λάθους ε, και πόσα κονδύλια δεν θα έπρεπε να έχουν εκταμιευθεί, αυτό θα το γνωρίζουμε με απόλυτη σαφήνεια μόνο εφόσον έχουν ολοκληρωθεί τα προγράμματα. Πράγματι είναι αλήθεια ότι ε, είναι υψηλό το ποσοστό του λάθους. Το 11% των κονδυλίων δεν θα έπρεπε να έχει εκταμιευθεί. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Είναι αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή αυτή είναι η κατάσταση. Κατά τα άλλα, όσον αφορά το ερώτημα σχετικά με την ποιότητα των ε, ελέγχων των λογιστικών ε, πρέπει να σα πω ότι το Συμβουλίο λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη του αυτού του ελέγχου, όπω επίση και την, ε, το συμπέρασμα, το πόρισμα του ε, ελεγκτικού συνεδρίου. Φαίνεται λοιπόν ότι δεν υπάρχει απόλυτη αξιοπιστία. Παρόλα αυτά, εμείς είμαστε πεπισμένοι ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καταβάλουν ε, πράγματι μεγάλη προσπάθεια και εγώ είμαι ακράδαντα πεπισμένος για το ότι στο μέλλον η έλεγχη αυτή των λογιστικών θα προσφέρουν πάρα πολλές δυνατότητες σε εθνικό επίπεδο. Υπάρχουν οι αποκαλούμενες πολιτικές δηλώσεις. Αυτό το έχουν αποφασίσει ορισμένα κράτη-μέλη. Και το Συμβούλιο δεν πιστεύει ότι αυτό πρέπει να αναχθεί σε επίπεδο αρχής. Το Συμβούλιο πιστεύει πολύ περισσότερο ότι θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα περισσότερη λογιστική έλεγχη. Ποιο είναι εκείνο που ρωτήσατε θα πρέπει να ορίσει το ποσοστό ε, ανοχής λαθών. Επ' αυτό το Συμβούλιο δεν τοποθετήθηκε και πρέπει να σας πω και εγώ δεν είμαι εξουσιοδοτημένος να τοποθετηθώ πάνω σε αυτό το ερώτημα γιατί δεν υπάρχει κατ' ουσίαν Βεβαίως μπορώ να σας πω την καθαρά προσωπική μου άποψη και αυτό πρέπει να το εκλάβετε όπως σας το λέω την άποψη του ε, Τσέχου Υπουργού Οικονομικών. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι εκείνος που ελέγχεται δεν θα πρέπει να ορίζει μόνος του το ποσοστό ανοχής λάθους, αλλά το ποσοστό αυτό θα πρέπει να γίνεται, να ορίζεται από τον ελεγκτή. Βεβαίως ενδέχεται μετά από εκτενή συζήτηση ε, να αλλάξει το ποσοστό και αυτό βέβαια θα εξαρτάται από τη συμφωνία που θα προκύπτει ανάμεσα στο ε, Συμβούλιο, την ε, Κομισιόν και το καθεξής. Οι ε, εθνικές αρχές είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένες, πάντως εγώ δεν πιστεύω ότι μπορούμε να επιτύχουμε συμφωνία, απόλυτη συμφωνία όσον αφορά την εφαρμοστέα μέθοδο. Γιατί ε, σε πάρα πολλά κράτη το Σύνταγμα είναι εκείνο που καθορίζει τη θέση που πρέπει να ε, ληφθεί και δεν μπορεί κανείς να επέμβει ούτε καν το ελεγκτικό συνέδριο. Βεβαίως ε, αυτό πρέπει να συζητηθεί εκτενώς. Όλοι μας οφείλουμε να παρακολουθήσουμε αυτά τα θέματα στις ε, πατρίδες μας και να ε, δώσουμε τις απαραίτητες λεπτομέρειες ε, στις ελεγκτικές αρχές. Πάντως, όπως σας είπα και προηγουμένως, υπάρχουν αυτά τα προπύρια, θα έλεγα, ελέγχου και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε σχεδόν τίποτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ε, θα ήθελα τώρα να μου επιτρέψει να δώσω το λόγο στο ελεγκτικό συνέδριο. Ίσως ε, ε, να αισθάνεστε κι εσείς ότι αμφισβητούνται οι γνώσεις σας το κατά πόσο είναι σημαντικό το 11% ή όχι ε, ίσως λοιπόν από ε, αυτού ε, μπορείτε κι εσείς να υπερασπιστείτε τη θέση σας. Θα σήμουν και ευγνώμων γιατί αυτό το χρειαζόμαστε για την απαλλογή. Δηλαδή τα αποτελέσματα στα οποία καταλήξατε έχουν κάποια διάρκεια, κάποια συνέπεια. Γιατί αλλιώς θα πρέπει να δώσουμε το λόγο στο Συμβούλιο. Κύριε Μπονίτσι, θέλετε να λάβετε εσείς το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Με ενδιαφέρε πολύ το ψήφισμα του Συμβουλίου. Το διάβασα μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι πιο προσεκτικό στη διατύπωσή του από αυτά που άκουσα. Το 11% που αναφέρεται ήπια, δεν ξέρω αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα κατανόησης ή όχι. Να εξηγήσω, το 11% είναι το χαμηλότερο επίπεδο σφάλματος. Δεν είναι το πιθανότερο επίπεδο σφάλματος, το σφάλματος που είναι φυσικά μεγαλύτερο. Λοιπόν, το μικρότερο ποσοστό σφάλματος που έχουμε αποφασίσει, όχι με 100% εμπιστοσύνη, διότι αυτό είναι ανέφικτο, αλλά με 95% εμπιστοσύνη. Είμαστε 95% λοιπόν σίγουροι ότι τουλάχιστον 11% δεν θα πρέπει να έχει πληρωθεί. Πέρσι ήταν 12%. Παρόμοιο φάσμα και πριν. Παρόμοιο ποσοστό. Επί σειρά ετών η εικόνα είναι παρόμοια που διαφαίνεται. Το ψήφισμα του Συμβουλίου σωστά αναφέρει ότι είναι και το θέμα του πολιετούς χαρακτήρα. Πράγματι. Το θέμα αυτό όμως δεν θα πρέπει να είναι θεωρητικό απλώς, αλλά πρέπει να ποσοτικοποιηθεί Δυστυχώς όμως δεν έχουμε τέτοια ποσοτικοποίηση. Εξετάζοντας το παρελθόν και την ολοκλήρωση των προγραμμάτων και το κλείσιμό τους, βλέπουμε ότι και πάλι η εντύπωση που αποκομίζουμε δεν είναι πολύ ξεκάθαρη και σημαντική. Η συνθήκη προβλέπει να διεξάγεται αυτή η διαδικασία ΙΟΣ και υπάρχει κάποιο στοιχείο πολιετούς χαρακτήρα της διαδικασίας. Το 11% όμως είναι αποτέλεσμα των αναλύσεών μας. Είναι το χαμηλότερο ποσοστό σφάλματος, αλλά όχι το πιθανότερο ποσοστό. Λέμε ότι είναι τουλάχιστον αυτό το ποσοστό για το οποίο είμαστε 95% σίγουροι. Στη δική μου γλώσσα, ε, τι να πω, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν είναι κόκοσά μου, δεν είναι κάτι απειροελάχιστο. Ίσως κάποιος μπορεί να δει μακροπρόθεσμα ποιες θα είναι εξελίξεις, Κάποιος μισμός οικονομολόγος είπε ότι μακροπρόθεσμα όλοι είμαστε νεκροί δυστυχώς. Άρα θα ήταν καλό να συλλέξουμε περισσότερες πληροφορίες και νομίζω ότι είναι δυνατό κάτι τέτοιο. Από τη μελλοντική προγραμματική περίοδο, ίσως πληροφορίες που θα έρθουν από τα κράτη-μέλη. Τώρα όμως αυτό δεν είναι επιχείρημα για να απορρίψει τα αποτελέσματά μας. Είμαστε πάντα ανοιχτοί. Μπορούμε να πιστούμε. Και ως ελεγκτές είμαστε ανοιχτοί σε στοιχεία. Το πρόβλημα είναι τα στοιχεία όμως. Ευχαριστώ. Ο Προεδρεύων θα λάβει αμέσως το λόγο, αλλά νομίζω ότι για μας ε, που είμαστε αρμόδις φορέας όλα αυτά που λέμε είναι σημαντικό. Δηλαδή το 11% στο οποίο καταλήξατε εσείς είναι κάτι το απλά γενικό αλλά έχει, μήπως έχει ουσία. Το Συμβούλιο και παραθέτω λέει ότι αυτή η εκτίμηση πρέπει να αντιμετωπιστεί cum granum salis. Ε, τι λέει αυτό, τίποτα δεν λέει. Ε, εγώ επαναλαμβάνω, επιμένετε σε αυτούς τους αριθμούς. Ελπίζω ναι, γιατί εσείς το προτείνατε και καταλήξετε σε αυτό και το Συμβούλιο λέει πολύ προσεκτικά. Τέλο πάντων, θα λάβει τώρα το λόγο το Συμβουλίο. Ελπίζω όμω όσον αφορά αυτό το θέμα να καταλήξουμε κάπου. Σα ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε. Στο ερώτημά σας ε, αναφέρατε ότι εγώ αμφισβήτησα ε, την τοποθέτηση του ελεγκτικού συνεδρίου. Αλλά δεν ισχύει αυτό. Εγώ δεν έχω κανένα λόγο να το κάνω αυτό. Το ελεγκτικό ε, συνέδριο ε, ακολούθησε την πεπατημένη. Και εγώ απλά επισήμανα την ερμηνεία του ποσοστού του 11%. Γιατί το ελεγκτικό συνέδριο δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο παρά να ελέγξει το 2007 τα προγράμματα που είχαν πολιετή χαρακτήρα. Δηλαδή, Δεν μπορεί κανείς ε, να συμπεραίνει από αυτό ότι αμφισβητούμε. Αυτή απλά είναι η αξιολόγηση ε, της μίας πλευράς. Στην περίπτωση των ε, πολιτών προγραμμάτων και δεν είμαι 100% σίγουρος κατά πόσον ε, θα πρέπει κανείς να συγκρίνει και την εμπειρία από τα προηγούμενα έτη. Νομίζω μάλιστα ότι δεν είναι καν δυνατόν να γίνει αυτή η σύγκριση. Γιατί το 2007 είναι η έναρξη μιας νέας περίοδου με νέα νομοθετικά μέτρα, νέους κανόνες. Εγώ λοιπόν θα δίσταζα ασυλλόγιστα να κάνω αυτή τη σύγκριση διότι παλαιότερα υπήρχε ισχύει υψηλότερο ποσοστό λάθους από αυτό που ισχύει τώρα. Την απόλυτη σιγουριά θα μπορέσουμε να την αποκομίσουμε αργότερα και γι' αυτό το λόγο εγώ θα ήθελα να σε επισημάνω και ένα κίνδυνο που υπάρχει εφόσον προσπαθήσουμε να ισχυριστούμε ότι το 11% των κονδυλίων δεν θα έπρεπε να έχει εκταμιευθεί ποτέ. Όποιος το λέει αυτό εκφράζει και δυσπιστία απέναντι στο ελεγκτικό συνέδριο. Εγώ δεν θα το έκανα ποτέ αυτό. Νομίζω ότι δεν πρέπει να αναφέρουμε αυτό τον αριθμό σε σχέση με τα πολιτή προγράμματα παρότι ε, το πόρισμα είναι απόλυτα σαφές. Πρόεδρος, ε, όπως είπαμε, ε, πρώτα θα γίνουν οι συζητήσεις και μετά θα ξαναμιλήσετε. Τώρα ο κύριος Μποτόπουλος, ε, να ζητήσετε όμως το λόγο αν θέλετε και βεβαίως κύριε Προεδρεύοντα και το Ελληνικό Συνέδριο καλούνται να τοποθετηθούν. Παρακαλώ. Ο συνάδελφος κύριος Μποτόπουλος. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Υπουργέ για την ανάλυση και τις παρατηρήσεις. Δράτω με τις παρουσίες σας και δεν ξέρω αν θα μείνετε για όλη τη συνεδρίαση Δράτω με τις παρουσίασεις να σας θέσω ένα ερώτημα που άμεσα συνδέεται με τα όσα είπατε, αλλά εκπροσωπείτε το Συμβούλιο και γι' αυτό θα σας ρωτήσω ποια είναι η απόψή σας για κάτι που πολλοί θεωρούμε ότι είναι πρόβλημα όταν δίνουμε την απαλλαγή του Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο. Δηλαδή, μας λείπουν στοιχεία, έγγραφα, τα στοιχεία εκείνα που θα μας επιτρέψουν να κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Κυρίως στον τομέα της κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής άμυνας. Ποια είναι η άποψή σας που είστε εκπρόσωπος του Συμβουλίου. Η Τσεχική Προεδρία θα κάνει κάτι περί αυτού. Κοιτάξτε, μου είναι πολύ δύσκολο να μιλήσω γι' αυτό, γιατί έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει κανείς να τηρεί τις ε, συμφωνίες των κυρίων. Ε, Βεβαίω γνωρίζω πολύ καλά ότι εδώ υπάρχει συμφωνία κυρίων ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο όσον αφορά τον προϋπολογισμό και εμένα μου αρέσουν αυτές οι συμφωνίες κυρίων. Άρα δηλαδή, ε, παρότι σέβομαι απόλυτα ε, τις αρμοδιότητές σας, ε, τη δυνατότητά σας να λαμβάνετε αποφάσεις. Εγώ θα ήθελα να σας παραπέμψω σε αυτή τη συμφωνία κυρίων και επίσης και στις σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στον αποκαλούμενο μεγάλο προϋπολογισμό που διαχειρίζεται η Κομισιόν και αφετέρου τους ε, διοικητικούς προϋπολογισμούς ε, του ε, Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. που βέβαια προφανώς και το τελευταίο ευρώ παίζει κάποιο ρόλο. Εδώ μιλάμε για διαφορετικά μεγέθη στη δεύτερη περίπτωση. Ε, γιατί στη δεύτερη περίπτωση ακριβώς επειδή τα μεγέθη είναι διαφορετικά το πρόβλημα είναι και πιο σχετικό. Ε, γνωρίζω επίσης ότι τα τελευταία χρόνια ο εκπρόσωπος ε, του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου είχε κάποια σχέση, ε, συγγνώμη, συνάντηση με τα μέλη του Κοινοβουλίου για θέματα που έχουν σχέση με την απαλλαγή και θεωρώ ότι ε, φέτος δεν θα λάβει χώρα αυτή η συζήτηση, δεν έγινε με πάση περιπτώσει, παρότι κατεβλήθησαν σχετικές ε, προσπάθειες. Τώρα το τι σκέφτομαι εγώ γι' αυτό, εγώ ε, πιστεύω ότι είναι καλό σε οποιαδήποτε περίπτωση να γίνονται συζητήσεις και συναντήσεις, να ανταλλάσσει κανείς ε, απόψεις και εμπειρίες. Έτσι λοιπόν, εγώ ε, σας παρουσίασα τη σύσταση του Συμβουλίου για την απαλλαγή του προϋπολογισμού της Κομισιόν. Εγώ θεωρώ ότι ο προϋπολογισμός της Κομισιόν είναι εντάξει. Διορθώνει ο προϋπολογισμός του Συμβουλίου είναι εντάξει. Κυρία Κρέσλε, κύριε Υπουργέ, ε, είναι πάντα δύσκολο να συζητήσει κανείς με τον εκπρόσωπο του ε, Συμβουλίου, αλλά τελικά ε, θεωρώ ότι ε, το Συμβούλιο όσον αφορά αυτά τα στοιχεία καλύτερα να τα ανεβάσει σε κομική επιθεώρηση γιατί έχουν κομική αξία. Με την εξή έννοια ότι για πολλωστή φορά δεν υπάρχει δήλωση αξιοπιστίας του χρόνου θα κάνουμε μάλιστα και γιορτή, θα το γιορτάσουμε επί 15 συνεχεία γιατί δεν θα έχουμε δήλωση εξοπιστία. θα είναι επέτειο. επαιτειακή ημερομηνία και φαντάζομαι ότι δεν θα παραμείνουμε στη 15η αλλά θα φτάσουμε και στην 20η επέτειο. Αλλά ξέρετε κάτι, α αφήσουμε τα αστεία, το κοινοβούλιο σιγά σιγά και εκνευρίζεται ε, διότι από ό,τι φαίνεται το Συμβούλιο ούτε καν ενοχλείται από τι διαπιστώσει. Κοιτάξτε, ε, βέβαια πρόβλημα σκέλος του προβλήματος είναι και τα κρατη Και όσο το Συμβούλιο προσποιείται ότι πρόκειται για ε, κάτι το αφηρημένο χωρίς να επισημαίνει ότι πρόκειται για κράτη-μέλη ε, τότε δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτόν τον τρόπο. Τι θα γίνει τελικά. Εμείς ε, εντοπίσαμε τα κράτη-μέλη που δημιουργούν πρόβλημα. Κατά την περίοδο 2000-2006 στα διαρθρωτικα ταμεια ταμεία είχαμε τρία-τέσσερα κράτη ε, τα οποία ε, σωρευτικά διέπραξαν το 95% των λαθών στα διαρθρωτικά ταμεία. Μιλάμε δηλαδή ε, για τα υπόλοιπα κράτη, τα 21, που αν εγώ ήμουν ένα από αυτά θα επέμενα να είναι όλοι ίσοι. Δηλαδή, όσον αφορά τη στρατηγική που ακολουθείτε για να εντοπιστούν τα λάθη, αυτή τη στρατηγική του Συμβουλίου εγώ δεν την ε, κατανοώ. Και τελικά όσον αφορά την ανοχή, εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Εσείς ε, λέτε ότι θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε και εντάξει θα το πράξουμε αυτό. Αλλά στη τελική ανάλυση και εσείς είστε ο άλλος βραχίωνας ε, της δημοσιονομικής πολιτικής. Ποια είναι η δική σας η θέση από αυτού, τι πιστεύει το Συμβούλιο. Θα ήθελα να θίξω και το θέμα της ε, Βουλγαρίας και της ε, Ρουμανίας. Σας υπενθυμίζω ότι εδώ πρόκειται για δύο κρατημέλη που προσεχώρησαν το 2007. Εν τω μεταξύ στη Βουλγαρία παγώσαμε το 1 τρίτο των ενισχύσεων και το Συμβούλιο δεν λέει τίποτα γι' αυτό. Ε, ως ε, ε, φορολογούμενοι και ευρωβουλευτήνα πρέπει να σας πω ότι εγώ είμαι παντελώς δυσαρεστημένη με τον τρόπο με τον οποίο το Συμβούλιο αντιμετωπίζει τα δικά του τα προβλήματα. Αυτό το πρόβλημα επήγει και μόνο εσείς ε, μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα σε συνεργασία με την Κομισιόν. Εμείς ε, βεβαίως να κάνουμε προτάσεις αλλά θα ήταν ιδιαίτερα θετικό εάν το Συμβούλιο, δεν είναι προσωπικό το θέμα, δεν είναι για σας, το Συμβούλιο, εάν το Συμβούλιο έδειχνε μια μεγαλύτερη προσπάθεια και μεγαλύτερη σοβαρότητα σας παρακαλώ παρακαλώ πάρα πολύ στη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ ε, για αυτήν την ε, ανοιχτή σας ε, τοποθέτηση. Αρχικά είπατε ότι για έναν εκπρόσωπο του Συμβουλίου η θέση του είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη επί της ουσίας, κυρίως διότι εγώ δεν είχα αρκετό καιρό για να παρακολουθήσω τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Παρ' όλα αυτά βέβαια πρέπει να σας πω ότι εδώ ανάμεσά σας αισθάνομαι πολύ καλά και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Κοιτάξτε, στην ομιλία μου εισαγωγικά Είπα ότι διαπιστώνεται βελτίωση κυρίως όσον αφορά τα συστήματα ελέγχου και ίσως να μην το τόνισα επαρκώς αλλά ανέφερα στην εισήγησή μου ότι το υψηλό ποσοστό λάθους ε, κυρίως ε, στα διαρθρωτικά ταμεία στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης όλα αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν με απλούστευση των ε, κανονισμών. Όταν είναι δύσκολοι κανονισμοί αυξάνεται το ποσοστό του λάθους. Γι' αυτό λοιπόν εμείς ως Συμβούλιο θα θέλαμε να καλέσουμε την Κομισιό να απλουστεύσει τους κανόνες. Ως ε, κράτη-μέλη προσπαθούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα της ε, διαχείρισης και τη δική μας την ποιότητα των ελεγκτών. Τα κράτη-μέλη είναι εκείνα τα οποία υποβάλλουν τις ετήσιες ε, συστάσεις ε, Το θέμα του κινδύνου δεν συζητήθηκε ακόμα στο Συμβούλιο και ελπίζω να τοποθετηθεί επ' αυτού ο διάδοχός μου. Η συζήτηση έχει προγραμματιστεί για την Άνοιξη. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας έκανα να χαμογελάσετε, αλλά πρέπει να σας πω ότι δεν είμαι σε θέση να σας ε, παρουσιάσω ε, μία ε, θέση οριστική. Η τελική θέση του Συμβουλίου θα προκύψει την Άνοιξη. Άρα δηλαδή για άλλη μια φορά σας ζητώ συγγνώμη η συνάδελφός μου μου επισημαίνει ότι κάνατε άλλη μια ερώτηση που αφορά στη Βουλγαρία. Εδώ πρέπει να σας πω ότι η Κομισιόν έκανε τη δουλειά της πολύ σωστά, είχε κάποιες αμφιβολίες, γι' αυτό λοιπόν ε, ανέστηλε απάραυτα την εκταμείευση των κονδυλίων διότι διαπίστωσε ότι δεν διεξάγονται οι απαραίτητοι έλεγχοι. Ο Μούλντερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω πολύ καλά τη χώρα σας, αλλά σαν υπουργό Οικονομικών θα ήσασταν σε θέση να έχετε 14, σε 14 διαδοχικά χρόνια αρνητική άποψη και γνωμοδότηση του ελεκτικού συνεδρίου και να εξακολουθείτε να βασίζεστε στην υποστήριξη του Τσεχικού Κοινοβουλίου για την εκτέλεση των καθηκόντων σας. Κυρίως όταν βλέπετε ότι η βελτίωση προχωρά με ρυθμούς πολύ αργούς. Ποια θα ήταν η στάση σε μια αξιότιμη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Πώς μπορείτε να πείσετε τους ευρωπαϊκούς λαούς ότι 14 διδυχικά χρόνια από ό,τι ξέρετε με μία διαφωνία μόνο δίνεται απαλλαγή στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στα πλούσια κράτη-μέλη πώς θα τα εξηγήσετε να δώσουν πίσω τους πώς περιφερειακά ταμεία. Όταν είναι πολύ κακή η χρήση των ποσών. Δεν ξέρω ποιο είναι το ποσοστό σφάλματος στην Τσεχία, αλλά 11% είναι το ελάχιστο, μπορεί να είναι και πάνω από το 11% το σφάλμα. Απαντώντας στο ερώτημα του κυρίου Βοτόπουλου, αναφερθήκατε συμφωνία κυρίων μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Η συμφωνία κυρίων είναι μεταξύ μερών που εμπιστεύονται το ένα το άλλο. Λόγω τιμής θα μπορούσατε να πείτε ότι δεν έχει κρυφό προϋπολογισμό στο Συμβούλιο για την ΚΕΠΑ και ότι όλες οι δαπάνες πηγαίνουν για διοικητικούς σκοπούς και μόνο. Ο κύριος Νομίζω ότι αυτή η κατάσταση θλίβει όλους μας. Θα ήταν λοιπόν λάθος να μην ε, διαπιστώσουμε ότι η κατάσταση αργά αλλά σταθερά βελτιώνεται. Ακριβώς διότι δεν πρόκειται για ένα και μόνο κράτος μέλος, αλλά για το ότι εδώ ε, συνεργάζονται 27 κράτη και πρέπει όλοι να συμφωνήσουν για το ποσοστό του λάθους. Για να γίνει αυτό ε, πρέπει να υπάρξει τουλάχιστον ειδική ε, πλειοψηφία. Τώρα είπατε τι θα ε, γινόταν στη δική μας τη χώρα αν επί 14 συναπτά έτη και ούτω καθεξής. Ε, κοίταξτε, εντωμεταξύ όμως ο υπουργό θάλαζε αρκετές φορές αυτά τα 14 χρόνια. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο μπορεί κανείς υποθετικά έστω να κάνει τέτοιο ερώτημα. Δεν ξέρω κατά πόσο έστω και υποθετικά μπορεί και να συγκρίνει την κατάσταση ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει κανείς να καταλήξει κάποια στιγμή σε συμφωνία. Νομίζω λοιπόν ότι όλοι πρέπει να αγωνιστούμε έτσι ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση. Συζητάμε για, το, ε, για την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Υπάρχουν ε, διαβουλεύσεις και όλα αυτά είναι καθορισμένα στο πλαίσιο της διοργανικής ε, συμφωνίας. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει η συμφωνία. Εγώ ε, σέβομαι αυτή τη συμφωνία και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι ε, ο προπολογισμό του Συμβουλίου ε, περιλαμβάνει μόνο διοικητικές ε, δαπάνες Εγώ λοιπόν πραγματικά δεν έχω καμία άλλη ενημέρωση και ως εκ τούτου μπορώ να σας ορκιστώ ότι και κανείς άλλος ότι δεν έχω πληροφορίες που να δείχνουν ή υπονοούν ότι υπάρχουν κάποια μυστικά κονδύλια. Ευχαριστούμε πολύ. Ο εισηγητής, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Εσείς είστε και εισηγητής σε αυτό το θέμα. Κύριε Υπουργέ, αναφερθήκατε στο θέμα της Συμφωνίας Κυρίων. και νομίζω ότι θα έπρεπε να το συζητήσουμε αυτό αργότερα. Επιτρέψτε μου όμως να θέσω δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις όσον αφορά τη Συμφωνία Κυρίων. Πρώτο ερώτημα. Αν αυτή η συμφωνία πραγματικά υπάρχει και ισχύει, συμφωνείτε να αποτελέσει τμήμα του κεκτημένου στο οποίο συμμορφωνόμαστε, μάλλον συμφώνησαν τα κάτι μέλη όπως χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν συμφωνίες που έχουν μια ισχύ συγκεκριμένη και οι χώρες που προσχωρούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το γνωρίζουν. Είναι κάποιε χώρε που είναι μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1975. Εσεί, η δική σα χώρα μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσφατα και μετά το 1979. Αυτή η συμφωνία κυρίων, αυτή η συμφωνία αποτελεί τμήμα της συμφωνίας που συνήψατε όταν προσχωρήσατε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτο ερώτημα αυτό. Το δεύτερο ερώτημα που έχω να σας θέσω. Όταν ο ίδιος κύριε Υπουργέ αναφέρεστε σε αυτή τη συμφωνία κυρίων, ποια παράγραφο αυτής της συμφωνίας κυρίων καλύπτει την ε, απαλλαγή που χορηγείται στο Συμβούλιο και που αφορά το θέμα της ΚΕΠΑ. Μελέτησα το θέμα και δεν μπόρεσα να βρω αυτή την παράγραφο. Θα ήθελα λοιπόν να μου δώσετε κάποια στοιχεία, να μας πείτε πού μέσα σε αυτή τη συμφωνία μπορούμε να βρούμε την παράγραφο τη σχετική που μεσα αυτη τη συμφωνια μπορουμε να βρουμε την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια Ευρωπαϊκής Ενώσεως και που αναφέρεται εκεί απαλλαγή στο Συμβούλιο. Κύριε Υπουργέ. Pane Κοιτάξτε, έχετε δίκιο. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα η οποία ε, προσεχώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004. Έτσι λοιπόν, έλαβε σάρκα και οστά ε, το όνειρό μας που εγώ ε, τον ονειρευόμουν την εποχή του κομμουνισμού. Τότε που δεν είδε μπορούσα να φανταστώ ότι θα βρισκόμουν κάποια στιγμή εδώ σε αυτήν την αίθουσα και θα μπορούσα να σας απευθύνω το λόγο. Ε, γι' αυτό λοιπόν εγώ λαμβάνω πραγματικά υπόψη μου όλες τις συμφωνίες και τις συμφωνίες ε, κυρίων και το κοινοτικό και εκτιμένο ε, και όλες τις άλλες ε, συμφωνίες που κάθε μία από αυτές έχει υπέρ και κατά. Όλα αυτά τα παίρνω πολύ σοβαρά υπόψη μου. Και είμαι ακράδαντα πεπισμένος ότι η διοργανική συμφωνία καλύπτει όλα αυτά. Θα ήθελα όμως να σας επισημάνω ότι η δική μου η εντολή που έχω είναι ε, να σας ε, παρουσιάσω τις ε, συστάσεις για την απαλλαγή της Κομισιόν, όχι του Συμβουλίου. Εκτιμώ ιδιαίτερα όλες τις ερωτήσεις που μου υποβάλλετε και πραγματικά προσπαθώ να απαντήσω. Όμως θεωρώ ότι η συζήτηση που κάνουμε εδώ δεν αφορά τα θέματα για τα οποία εγώ είμαι αρμόδιος εντάξει, υπάρχουν ε, κάποιοι συνάδελφοι που το έχουν θίξει το θέμα. Παρακαλώ, έχετε και πάλι το λόγο. Αν μου επιτρέπετε, αυτή τη στιγμή ήθελα να σας ενημερώσω ότι συνεδριάζουν τα Εθνικά Κοινοβούλια με τον κύριο Πέτερινγκ και εντός ολίγου πρέπει να πάω και εγώ εκεί για να τοποθετηθώ στο θέμα της ε, παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Ε, γι' αυτό λοιπόν ε, πρέπει να σας ζητήσω συγγνώμη επειδή η συζήτηση δεν αφορά πλέον την απαλλαγή της Κομισιόν. Νομίζω ότι εξάντλησα τις δυνατότητες που έχω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ιδιαίτερα επικοδομητική συζήτηση και εδώ θα μου επιτρέψετε και να επισημάνω το πόσο σημαντικές είναι οι κοινέ μας ε, προσπάθειες, δηλαδή ε, να υπάρχει χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Βεβαίως και υπάρχουν πράγματα ε, τα οποία μας ταλαιπωρούν, παρακολουθώντας όμως την τάση καταλήγουμε στο ότι υπάρχει βελτίωση. Με κάθε σεβασμό λοιπόν προς τις ε, αποφάσεις επιτρέψτε μου να σας καταθέσω και εγώ τη σύσταση του Συμβουλίου για να αποφανθείτε επ' αυτής. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα το ότι μπόρεσα σήμερα να σε απευθύνω το λόγο. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Προεδρεύοντα και σας ευχόμαστε καλή δουλειά, καλή τύχη και θα λάβουμε υπόψη μας τις ε, συστάσεις σας. Υπάρχει κάποιος εδώ από το Συμβούλιο ή να το διαλύσουμε, λέει ο Πρόεδρος. Λιγάκι περίεργο αυτό που συμβαίνει. Ε, εγώ το βρίσκω πάρα πολύ περίεργο ότι δεν ε, μένει κανείς από τη γραμματεία του Συμβουλίου όταν φεύγει ο Προεδρεύων. Τέλος πάντων, ίσως να επανέλθουν αργότερα. Κύριε Κάμουρη, ζητήσατε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα περισσότερα ερωτήματα ετέθησαν. Και ο συνήθως παίρνουμε απαντήσεις που δείχνουν ότι δεν υπάρχει πραγματική προθυμία να γίνουν τα δύο πράγματα που χρειάζονται. Πρώτον, διευκρίνηση και απλούστευση των μεθόδων εργασίας των κανόνων και δεύτερον, να εφαρμοστεί μια αποτελεσματική δίκηση. Θεωρώ ότι το τελευταίο ερώτημα του κυρίου Μούλτερ δεν απαντήθηκε. Και διερωτώ με μήπως θα μπορούσαμε να θέσουμε γραπτός το ερώτημα. Είναι σημαντικό ερώτημα, ουσιαστικό ανεξάρτητα βλέπετε από το πώς βλέπουμε το ρόλο μας και τις ευθύνες μας, είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε επακριβώς τι περιέχεται και τι δεν περιέχεται στον προπολογισμό, τι βλέπουμε και τι δεν μπορούμε να δούμε. Άρα, κύριε Πρόεδρε, από εσά εξαρτάται, το αφήνω σε εσά να στείλετε το αναγκαίο γραπτό ερώτημα για να λάβουμε απάντηση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, νομίζω ότι εδώ υπάρχουν ε, κάποια ερωτήματα, κυρίως όσον αφορά την ε, Συμφωνία Κυρίων. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά, το είπε και η κυρία Κρέσλε, ότι για 14η φορά τα κράτη-μέλη λένε ότι εντάξει όλα καλά και κάποια στιγμή θα πούνε, μα τι γίνεται τελικά στι Βρυξέλλε. Νομίζω ότι αυτή την ευθύνη πρέπει να την αναλάβουμε. Αυτή είναι η δουλειά μα. Ε, Κανεί δεν μπορεί να μα βοηθήσει. Ε, και καταλαβαίνετε ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να το παρουσιάσουμε και στου εκλογεί μα. Μπορούμε λοιπόν να κλείσουμε αυτό το θέμα. Γιατί σα λέω, είναι σημαντικό ε, και θα ήθελα να τα πούμε όλα αυτά με απόλυτη σαφήνεια στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και στο ελεγκτικό συνέδριο. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε ότι οι απόψεις πρέπει να ερμηνεύονται με ε, προσοχή. Αυτό είναι εκείνο που αναφέρεται στη συμφωνία. Και βεβαίως ε, σε τελική ανάλυση αυτό το κρίνει ο εκάστοτε εισηγητής. Πάντως Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει σαφήνεια όσον αφορά αυτό το θέμα γιατί αλλιώς ε, δεν μπορούμε να καταρτήσουμε έκθεση. Κοιτάξτε, για την επόμενη συνάντησή μας με το Συμβούλιο, εγώ ε, λέω να πούμε ότι κοιτάξτε το θέμα αυτό έχει κλείσει. Γιατί ε, το γεγονός ότι τώρα αυτοί σηκώθηκαν και έφυγαν, ειλικρινά σας λέω τώρα αυτό τι να πω, δεν είναι σωστό. Το ελάχιστο που μπορώ να πω. Ε, θα επανέλθουμε στο θέμα, πολύ σωστά το είπατε. Τι να κάνουμε, άνθρωποι είμαστε όλοι, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Πάμε στο επόμενο σημείο, στο υπαριθμό 7, απαλλαγή του 2007. Ε, ο κύριος Οντί είναι το αρμόδιο μέλος και ε, έτσι λοιπόν ε, θα θέλαμε εδώ να καλωσορίσουμε και τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Κάλλας. Έχουμε εδώ και πάρα πολλά μέλη του Συμβουλίου που είναι αρμόδια για το θέμα αυτό. Πρώτα απ' όλα δίνω το λόγο στον κύριο Οντί. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια που τελειώσαμε με το προηγούμενο σημείο, αναφερόμενοι στην Προεδρία του Συμβουλίου και ο Υπουργός δεν απάντηση για το κατά πόσο θα είναι στην Ολομέλεια όταν θα συζητήσουμε την απαλλαγή. Θέλω να επιμείνω σε εσά, Πρόεδρε, να περάσετε το μήνυμα αυτό στο Συμβούλιο, ώστε στην Ολομέλεια να μα κάνουν τη χάρη να βρίσκονται στα έδρανα του Συμβουλίου. Για την παρουσίαση τώρα της ε, απαλλαγής. Θέλω να ευχαριστήσω τον Αντιπρόεδρο τον κύριο Κάλλας για το ότι ήταν πάντα διαθέσιμος, για τις απαντήσεις που έδωσαν οι υπηρεσίε του στις ερωτήσεις μου και θέλω επίσης να ευχαριστήσω και το ελεγκτικό συνέδριο για όλες τις συνεδριάσεις που είχαμε μαζί, όπως επίσης να ευχαριστήσω και τους εισηγητές των πολιτικών ομάδων και την γραμματεία σας κύριε Πρόεδρε, κυρίως την κυρία Καστίγιο. Για άλλη μια φορά ευχαριστώ και τον προκάτοχό μου, τον κύριο Γιόγκερσεν, για τα έγγραφα για το 2006 που μου έδωσε και από τα οποία εμπνεύστηκα. Λοιπόν, περί πρόκειται, ξέρετε όλοι λίγο πολύ. Πρώτα απ' όλα έρχομαι στα οριζόντια ζητήματα. Όπως κύριε Κρεσλέτση και εγώ λυπάμαι που για 14η χρονιά έχουμε μια αρνητική δήλωση αξιοπιστίας. Διαπιστώνουμε βέβαια βελτίωση των συστημάτων ελέγχου, αλλά η βελτίωση αυτή δυστυχώς είναι πολύ αργή και ανεπαρκής. Χαίρομαι που στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου τα έσοδα και οι δαπάνες διοικητικέ δείχνουν, ε, καταδεικνύουν μάλλον τα λάθη που γίνονται. Για τους λογαριασμούς. Έχω βάλει μία σημείωση που είχα πει προφορικά αρχικά που λέει ότι οι διπόροι που παγιώνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά έχουν 58 εκατομμύρια ευρώ. Μου λένε ότι είναι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, τα διεθνή λογιστικά πρότυπα του δημοσίου τομέα. Όμως παρόλα αυτά εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το ψάξουμε περισσότερο και γι' αυτό και θα καταθέσω τροπολογία για τα 33 δις τα οποία οφείλουμε στο προσωπικό μας. Πιστεύω ότι δεν είναι λογικό να θεωρούμε ότι οι συντάξεις που χρωστάμε στο προσωπικό ε, παραμένουν ενώ έχουν πληρώσει εκείνοι ότι έπρεπε να πληρώσουν. Τα κράτη-μέλη όμως δεν τους δίνουν τα χρήματα αυτά. Θα επανέλθω. Κάτι άλλο που δεν καταλαβαίνω είναι για το χείρμα Γαλιλαίο. Η πολιτική συμφωνία υπάρχει για το δημόσιο τομέα, ήδη από το 2007, όμως τα λογιστικά δεν αναφέρεται. Θέλω λοιπόν να σας ζητήσω να μελετηθεί γιατί δεν έχουν συμπεριληφθεί τα ποσά ε, τη απουσία απόσβεσης. Όσον αφορά τώρα την νομιμότητα των ε, διαφόρων δραστηριοτήτων για τα εκτελεστικά όργανα δεν υπάρχει τίποτα το ιδιαίτερο, όμως για τις εισπράξεις θα τα διαβάσετε και για τις ε, εθνικές δηλώσεις αξιοπιστίας και τις ετήσιες ε, περιλήψεις. Το διάβημα είναι ορθό πιστεύω. Το είδαμε και πριν. Χρειάζεται ποιότητα και η ποιότητα διαφέρει κατά περίπτωση. Πράγμα το οποίο μας εμποδίζει να βγάλουμε σωστό συμπέρασμα όσον αφορά τον έλεγχο του κοινού ελέγχου που γίνεται. Για τις εθνικές δηλώσεις προτείνω να επαναλάβουμε το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να έχουμε τέτοιε εθνικέ δηλώσει αξιοπιστία. Λέω στην εκθεσή μου και το έχουμε συζητήσει μεταξύ συναδέρφων ότι υπάρχουν χώρε που υπογράφουν τέτοια δήλωση και άλλε που δεν υπογράφουν τέτοια δήλωση αξιοπιστία. Θέλω να ξέρω τη γνώμη των συναδέρφων. Εγώ λέω ότι υπάρχει η νομική βάση 248 όπου υπογραμμίζεται η τεχνική συνεργασία με το, ελεγκτικό, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και τις εθνικές αρχές και πρέπει να συμπεριλάβουμε και την ιδέα ότι στη διαδικασία απαλλαγή πρέπει να υπάρχει μια διαθεσμική, ένας διαθεσμικός μηχανισμός που θα ξανασυζητηθεί και θα αποφασιστεί και από τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια στη συνέχεια θα πηγαίνουν στις κυβερνήσεις βάσει, επαναλαμβάνω, κατάλληλης διαδικασίας απαλλαγής. Για το σύστημα ελέγχων. Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για το πρόγραμμα δράσης όσον αφορά τον εσωτερικό έλεγχο, τον ολοκληρωμένο. Όντως υπάρχει πρόοδος. Όμως ήρθε η στιγμή να γίνει και μία αξιολόγηση και σε τεχνικό επίπεδο αλλά και σε ηθικό επίπεδο. Γιατί πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι ο εσωτερικός αυτός έλεγχος είναι ανεξάρτητος τόσο ώστε να μπορεί να ληφθεί υπόψη στα διαβήματα τόσο ελέγχου του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου όσο και της επιμέρους ε, αξιολόγησης. Τώρα για το ανεκτό κίνδυνο σφάλματος. Εδώ δεν πιστεύω εγώ ότι είναι οι πολιτικοί εκείνοι οι οποίοι θα πρέπει να ανακατευθούν στην μεθοδολογία ελέγχου. Το ποσοστό ανεκτού κίνδυνου σφάλματος είναι κάτι που έχει να κάνει με την αξιολόγηση. Δεν είναι οι πολιτικές αρχές που πρέπει να καθορίζουν το ανεκτό κίνδυνο σφάλματος, αλλά οι αρχές ελέγχου. Και πρέπει εδώ πέρα να διευκρινίσουμε ποια είναι η σχέση ανάμεσα στον ανεκτό κίνδυνο σφάλματος που εφαρμόζεται στο σύστημα το ολοκληρωμένου εσωτερικού ελέγχου και το όριο εκείνο το οποίο χρησιμοποιείται από το ελεγκτικό συνέδριο. Γιατί πολλαπλασιάζοντας τα μέσα ελέγχου, καταλαβαίνετε ότι οι ευρωβουλευτές και οι πολίτες τελικά δεν θα καταλαβαίνουν πια τίποτα τι είναι αυτό το οποίο είναι αποδεκτό, ανεκτό, σημαντικό κλπ. Όλα αυτά είναι τεχνικά ζητήματα. Στο τέλος όμως έρχεται η ψηφοφορία του Κοινοβουλίου και η εκτίμηση που κάνουν οι πολίτες. Για τα επιμέρους τώρα θέματα, τα τομεακά. Γεωργία πρώτα απ' όλα. Εδώ προτείνουμε περισσότερη απλοποίηση. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Για τη συνοχή εδώ έχω βάλει μία παράγραφο με έναν προσωπικό προβληματισμό. 180 πληρωμές από 200.000 είναι κάτι που φτάνει ως δείγμα. Εδώ θα προτείνω τροπολογία να ξέρετε για να πω ότι εφαρμόζοντας την τεχνική αναθεώρηση στο ελεγκτικό συνέδριο φαίνεται ότι η τεχνική συνάδει με τις διεθνείς προδιαγραφές ελέγχου. Όσον αφορά την έρευνα και εδώ κάτι για τα πιστοποιητικά ελέγχου, τα οποία κοστίζουν πολλά χρήματα, χωρίς να έχουμε και απόλυτη εγγύηση. Για τον πολιτισμό και την παιδεία ζητάμε από την Επιτροπή Εναρμόνιση των δηλώσεων αξιοπιστίας εκ των προτέρων. Πάω γρήγορα γιατί νομίζω ότι όλοι την ξέρετε την έκθεση, δεν χρειάζεται να καθυστερήσω. Προτιμώ να ακούσω τις ερωτήσεις των συναδέρφων. Εξωτερικές δράσεις. Εδώ έχουμε πολλές ανησυχίες. Αναρωτιέμαι μήπως θα έπρεπε να διευκρινίσουμε όλες τις δομές παρέμβασής μας σε εξωτερικές δράσεις. Στα αναπτυξιακά ταμεία που να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται, γιατί μερικές φορές καταλήγουν να πρόκειται για διακυβερνητικές δράσεις και όχι για κοινοτικέ δράσεις. Τι περνάει από το ελεγκτικό συνέδριο, τι όχι. Εδώ δηλαδή υπάρχει ένα ολόκληρο σύνολο που πρέπει να ξεκαθαριστεί, να αποσαφινιστεί, για να μπορεί να γίνει καλύτερα και ο έλεγχος. Έρχομαι τώρα στις στην προταξιακή στρατηγική. Δεν χρειάζεται εδώ βέβαια να επαναλάβουμε τις ανησυχίες που έχουμε εκφράσει πολλές φορές στην Επιτροπή μας για τη Βουλγαρία πρώτα απ' όλα και τη Ρουμανία και το Κωσυφοπαίδιο. Αυτό όμως που κάνω εγώ είναι ότι ανανεώνω μία πρόταση που είχα κάνει παλιότερα, δηλαδή ζητάω να έχουμε παρέμβαση του Εθνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου του Κωσυφοπεδίου. Όταν πήγαμε για να εξετάσουμε τις παρεμβάσεις εκεί υπέρ αυτής της χώρας, ε, διαπιστώσαμε ότι χρειάζεται κάτι τέτοιο. Για τις διοικητικές δαπάνες τώρα. Τίποτα ιδιαίτερο. Για τις υποδομές της κοινότητας. Εδώ πάλι εκφράζω την ανησυχία μου για την Επιτροπή όσον αφορά την κοινοποίηση κάθε νέου σχεδίου υποδομών. Το κάνει, αλλά πιστεύω ότι οι πληροφορίες που μας δίνει θα πρέπει να είναι ακριβέστερες. Και ολοκληρώνω, Πρόεδρε, λέγοντας ότι δεν υπάρχει τίποτα ιδιαίτερο σε σχέση με τις ειδικές εκθέσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Εδώ έχω αντιγράψει copy-paste όλα όσα είχαν γράψει οι συνάδελφοι. Συνεπώς, προτείνω στο Κοινοβούλιο να ψηφίσει την απαλλαγή. Συγχρόνω όμως θέλω να πω στον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι έχω την αίσθηση ότι η σημερινή κατάσταση, και νομίζω ότι από αυτού συμφωνούν και οι συνάδελφοι, δεν είναι ικανοποιητική και πολύ θα ήθελα να τον ακούσω να μας πει στα τέλη της θητείας, εντάξει εδώ πρόκειται για την απαλλαγή 2007, αλλά καταλαβαίνετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κάνει μια συνολική αξιολόγηση για τον τρόπο με τον οποίο ε, εκτέλεσε την εντολή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ξεκίνησε από την υπόσχεση θετικής δάση. Μια λοιπόν καλή απάντηση, κύριε Αντιπρόεδρε, θα ήταν να μας πείτε πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα και ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε ώστε να είμαστε σε θέση να ελπίζουμε κάποια μέρα σε μια θετική δήλωση αξιοπιστίας, μια θετική τάση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σιγητά. Πράγματι, πίσω από τα λίγα λόγια που είπατε, κρύβεται πολλή δουλειά. Ο κύριος Αντιπρόεδρος, ο κύριος Κάλλας, παρακαλώ έχετε το λόγο. Κύριε Σιγητά, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την καλή και επικοδομητική έκθεση και την πρόταση να χορηγηθεί η απαλλαγή για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2007. Το σχέδιο εκθέσεως συμπεριλαμβάνει πολλές επικοδομητικές συστάσεις που αν υιοθετηθούν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει να τι δεχτεί και να τι εκτελέσει. Βεβαίω θα αποστείλουμε στον εισηγητή γραπτό σχόλια, αλλά επιτρέψτε μου ακροθυγώ να αναφερθώ σε σημεία όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαφορετική άποψη ή εκεί που το ψήφισμα χρήζει διευκρινήσεων. Η έκθεση προσδίδει μεγάλη προσοχή στου ανθρώπινου πόρου, στην πολιτική ανθρωπίνων πόρων και κτηρίων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι που αφασχολεί το ελεγκτικό συνέδριο. Αν δεν ήταν πολύ συνεπή ο έλεγχο του προσωπικού, είτε χρησιμοποιούνταν διαφορετικέ μέθοδοι. Η παράγραφο 121 συνεπώ, κατά την άποψή μα, πρέπει να διαγραφεί. Κινητικότητα του προσωπικού. Είναι μια καλή πολιτική, αλλά θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για ευαίσθητε θέσει και μόνο. Και αυτό δεν αναφέρεται στο 123, στο σημείο 123. Επίσης θα θέλαμε να καλέσουμε την Επιτροπή και τον εισηγητή να επανεξετάσουν είναι να διατυπώσουν τις παραγράφους 124, 125 και 127 που αφορούν την κτηριακή μας πολιτική. Πρέπει να πω ότι προσωπικώς επένδυσα πολλές προσπάθειες ούτως ώστε να γίνει καλύτερη, ο ευρωπαϊκός χώρος καλύτερη γειτονιά. Η πολιτική μας είναι διαφανής και με τις προτάσεις για τον προπολογισμό και για κάθε σημαντικό πρόγραμμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται πλήρως. Βεβαίω θα πρέπει να υπάρξει σαφή διοικητική αυτονομία και ευθύνη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα παρενέβαινε στα στη διαχείριση των κτηρίων των άλλων θεσμικών οργάνων ακόμα και είναι πρόσδεκτη μια συνεργασία. Επίση, θεωρώ ότι το κείμενο για τη διαχείριση των πόρων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία ίσω να είναι πολύ σκληρό. Στην προσχώρηση επεσήμανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σοβαρέ ανησυχίε σχετικά με την οικονομική διαχείριση. Η διαπίστευση δόθηκε αργότερα το 2007 και υπό συγκεκριμένου όρου. Μετά από αποστολέ που έγιναν ελέγχου το 2008, ανεστάλησαν οι χρηματοδοτήσει. Η Όλαφ τώρα συνεργάζεται στενά με την ε, Ρουμανία και τη Βουλγαρία και τι αρχέ των χωρών αυτών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιμένει επί τη δυνατότητα διαχειρίσεω των πόρων και επινομικών και δικαστικών μεταρρυθμίσεων. Συμφωνώ πλήρω ότι η κατάσταση δεν είναι ιδεώδη, αλλά έχω κάθε εμπιστοσύνη ότι τα οικονομικά συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω προστατεύτηκαν και αντλήσαμε μαθήματα για το μέλλον. Τώρα, όσον αφορά τι παραγράφου 5, 7, 8, δεν νομίζω ότι δικαιολογούνται απόλυτα. Η, η λογιστική πρακτική τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ευθυγραμμιστεί με τα λογιστικέ προδιαγραφέ τη διεθνή Τώρα σε μια σύσταση που δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε θα, να αναφερθώ στην παράγραφο 57 περί Γεωργίας ζητείται οι οικονομικές διορθώσεις να πρέπει να καταβάλλονται το τελικό, τελικό Αυτό θα παρεμπόδιζε το, το λογιστικό σύστημα και θα παρεμπόδιζε ε, την ανάκτηση πόρων του ευρωπαϊκού προπολογισμού. σε πολλά σημεία προτείνεται νέες υποχρεώσεις ενημέρωσης και υποβολής αναφορών για πληροφορίες που ήδη διαθέτουμε στο σημείο 33, 39, 67. Το σχέδιο εκθέσεως περί απαλλαγής ζητά καταλόγους των επιδόσεων των συστημάτων των κρατών μελών, αναφορά τους. Εγώ κατανοώ αυτή την ιδέα και την υποστηρίζω, αλλά νομίζω ότι καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος θα ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίζει η υποβολή αναφορών σχετικά με προβληματικούς τομούς στις αιτήσεις εκθέσεις δραστηριοτήτων των γενικών διευθύνσεών της. Βασίζονται σε κάθε κάτω μέλος οι εκθέσεις, διατίθεται στο Κοινοβούλιο και στο ευρύτερο κοινό κάθε χρόνο. Κύριε Ισηγητά, είναι σημαντικό αυτό που θέσατε. Στην παράγραφό σας 43 αναφέρεται Φέρεται το πώ μπορεί να επιτευχθεί θετική δήλωση εξοπιστίας μέσω μια διασκέψης που μπορεί να βασιστεί στη σύγκληση μεταξύ θεσμικών οργάνων και να βρούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Η Γερμανία ανέφερε ότι η διαδικασία διαδικασίας εξοπιστίας του 248 της συνθήκης ΕΟΚ δεν λειτουργεί και υποστηρίζει την άποψη του ελεκτικού συνεδρίου για τον εκτό κίνδυνο σε κάθε τομέα πολιτική. Θα πρέπει να γίνει συζήτηση εκθέτω το θέμα τη διασκέψη αυτή θα μπορούσε να βοηθήσει στι διαπραγματεύσει μου στο Συμβούλιο να έχω μια στεναρή υποστήριξη πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά για μία ακόμη φορά θα ήθελα να πω κάποια πράγματα, κάποια λόγια που πιθανότατα να μην έχω την εντολή να τα πω. Είπε και ο Υπουργό ότι δεν μπορεί να πει κάποια πράγματα για τα οποία δεν του έχει δοθεί εντολή. Να πω κι εγώ κάποιες σκέψεις μου για ένα σημαντικό θέμα, για τη δήλωση εξοπιστίας. Βεβαίως πρέπει να απαλλαγούμε από αυτήν και πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες ούτω ώστε να πετύχουμε τη θετική δήλωση εξοπιστίας. Κατά την άποψή μου υπάρχουν τρεις μεγάλες δυνατότητες. Πρώτη, να φύγει το μυστήριο από την όλη φράση. Ποια είναι η φράση αυτή. Το ελεκτικό συνέδριο δεν μπορεί να πει στο κοινό και σε εμά και σε εσά ότι όλες οι συναλλαγές είναι νόμιμες και κανονικές. Αυτό είναι ένα πόρισμα του ελεκτικού συνεδρίου που ερμηνεύεται ως τα πάντα να βαίνουν κακός και ότι σπαταλώνται πολλά χρήματα και ούτω καθεξής. Μυστήριο καλύπτει λοιπόν αυτή την φράση. Και είναι δυσνόητη. Και όλες οι συζητήσεις δείχνουν ότι έχουμε πετύχει πολλές βελτιώσεις. Τι δυνατότητες υπάρχουν να έρθει το πέπλο μυστηρίο από τη φράση, δεν ξέρω. Κάτι αναφέρεται, στη, συμπεριλαμβάνεται αυτό συνθήκη και εμείς δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε τροποποίησης των συνθήκων σε αυτή τη φάση. Το δεύτερο σημαντικό ζήτημα είναι, είναι το ανεκτό ποσοστό κινδύνου. Το ελεκτικό συνέδριο συνέβαλε τα μάλα στον τομέα αυτό. τους αυτά τα χρώματα σαν τα σήματα κυκλοφορίας που πάντα τα έχουμε υπόψη μας όταν συζητούμε. Τρίτον, τα, ταμεία, τα χρήματα του Ταμείου Συνοχής χρειάζονται ριζοσπαστική προσέγγιση. Δεν έχω εντολή να πω αυτά που λέω. Προσωπικές απόψεις εκφράζω. Παραδείγματο χάρη, αν τα ταμεία συνοχή διερθούν στα δύο, ένα κομμάτι πάει στι στοχότερε περιφέρειε τη Ευρωπαϊκή Ένωση που καθορίζονται από την Eurostat έτσι και είναι πλήρη ευθύνη των κρατών μελών, ποιοι κανόνε εφαρμόζονται, οι έλεγχοι που διεξάγονται κλπ. και οι δηλώσει που υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περιορθής διαχειρίσεως των πόρων και το άλλο τμήμα που το χειριζόμαστε σε κεντρικό επίπεδο. Χειριζόμαστε το πρόγραμμα σε κεντρικό επίπεδο. Μπορούμε να απορροφήσουμε τα μεγάλα προγράμματα. Συζητούνται προγράμματα υποδομής σε αυτή τη φάση. Τα χρειαζόμαστε. Ενεργειακά προγράμματα αναφέρονται. Και αυτά μπορούμε να τα διαχειριστούμε σε κεντρικό επίπεδο. Να μπορεί να αξιολογηθούν, να παρακολουθηθούν, να ελεγχθούν σε κεντρικό επίπεδο και είναι σαφέστατη εικόνα περί των αποτελεσμάτων του το τρόπο. Την τελευταία φορά που ήμουν εδώ και συζητούσαμε το θέμα των εκ... του κινδύνου, είχαμε πει ξεκινήσουμε μια συζήτηση ξεκινώντα από το κόστο των ελέγχων. Και επίσης και επί της αξιολογήσεως των πολιτικών αποτελεσμάτων, που είναι κάτι άκος περίπλοκο. Όπως σας είπα, αυτοσχεδιασμός ήταν τα τελευταία σχόλια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Αντιπρόεδρε. Μήπως υπάρχουν παρατηρήσεις εκ μέρους του ελεγκτικού συνεδρίου για αυτό το σχέδιο του εισηγητή. Ο κύριος Μπονίτσι, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το σχέδιο ψηφίσματος είναι λεπτομερές τατό. Άκρος επικοδομητικό. Πρέπει να εξεταστούν οι προτάσεις. Ήδη αναφέραμε κάποια σημεία στον εισηγητή. Θα υποβληθούν και άλλες τροπολογίες από ό,τι κατάλαβα. Θα βοηθούσε συζήτηση για τις 180 συναλλαγές. Αν αρκεί. Αυτό φορά τη μεθοδολογία. Η μεθοδολογία εξετάστηκε μικροσκοπικά, επανειλημμένως, σε μικροσκοπικό επίπεδο. Καλύτερο θα ήταν να εστιαστούμε περισσότερο όχι στο πώς φέρνει ο αγγελιοφόρος το μήνυμα, αλλά πώς θα βελτιώσουμε το τελικό αποτέλεσμα. Προσπάθησα να το εξηγήσω παρουσία του Υπουργού το ζήτημα. Το αποτέλεσμα που έχουμε είναι πολύ βάσιμο. Πολύ ισχυρό. Συνάδελφοι, όταν και εγώ και το συνέδριο λέμε ότι το χαμηλότερο ποσοστό, το ελάχιστο ποσοστό κινδύνου στατιστικό 95% σίγουρο χρησιμοποιούμε τώρα στατιστικές έννοιες δεν είναι συνηθισμένη διατύπωση σημαίνει ότι έχουμε πάνω από 11% σφάλμα. Ατυχώς αυτό το αποτέλεσμα υφίσταται και ταιριάζει και με τα αποτελέσματα προηγουμένων ετών. Ήταν πάλι πάνω από 180 συναλλαγές που εξετάστηκαν. Ίσως πρέπει να σιαστούμε λιγότερο στον τρόπο με τον οποίο ο αγγελιοφόρος παραδίδει το μήνυμα και περισσότερο να με το τι μπορεί να κάνουμε. Ο κύριος Κάλλας εδώ άνοιξε ενδιαφέρουσες διόδους. Διότι είναι ξεκάθαρο ότι για να βελτιωθούν τα πράγματα χρειάζεται επαναπροβληματισμός, εκ νέου ανάλυση του τομέα των διαθετικών ταμείων και όχι μόνον. Και κάποιοι άλλοι τομείς χρειάζονται ανάλυση καινούργια. Κυρίως πώς μπορούμε να επιφέρουμε βελτιώσεις ούτως ώστε εν τέλει τα χρήματα να δίνουν αποτελέσματα. Κάτι που θέλει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Να μην χρησιμοποιείτε τα χρήματα με λάθος τρόπο. Στο ελεκτικό συνέδριο επανειλημμένα τονίσαμε ότι χρειάζεται να εστιαστούμε περισσότερο στην απλούστευση. Να εστιαστούμε περισσότερο στο πώς όταν δημιουργούνται τα προγράμματα, όταν οργανώνονται, να προβλέπετε το κόστος των ελέγχων. Και το κόστος αυτό να είναι σε εύλογο επίπεδο. Και αν όχι, αν δεν γίνεται αυτό, ίσως πρέπει να επαναξεταστεί η δομή των πόρων. Αυτό είναι ένα καλό μήνυμα που το μέλλον. Αυτή είναι η σωστή προσέγγιση μελλοντική. Όσον αφορά για τα υπόλοιπα του ψηφίσματος της απαλλαγής, παρακολουθούμε προσεκτικότατα τη συζήτηση, ετοιμάσαμε κάποιες συστάσεις και ελπίζουμε να ληφθούν υπόψη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν ακούσαμε και ε, τις παρεμβάσεις των μελών. Ο κύριος ε, Γιούργινσεν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Όντι πρώτα απ' όλα, τον εισηγητή. Ήμουν στη θέση σας πέρυσι, οπότε ξέρω πολύ καλά τι τραβάτε. Και εκτιμάω ιδιαίτερα τη δουλειά σας. Εννοείται, εμεί στη σοσιαλιστική ομάδα έχουμε τις ίδιες ανησυχίες όπως και οι υπόλοιποι εδώ στην Επιτροπή μας ότι για άλλη μια φορά το ελεγκτικό συνέδριο δεν μπορεί να συστήσει μια θετική τάση. Και πιστεύω ότι για πολλούς λόγους φέτος τα πράγματα είναι κάπως περίπλοκα όσον αφορά αυτή τη διαδικασία. Γιατί τα τελευταία δύο χρόνια ιδιαίτερα πέρυσι, στην Επιτροπή μας μπορέσαμε να πιέσουμε την Επιτροπή και οι Επίτροποι ανέλαβαν κάποιες νέες πρωτοβουλίες οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ όταν τα αποτελέσματα δεν θα ήταν πια ορατά φέτος για τη φετινή μας έκθεση. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ενισχυτικά συμπεράσματα από το ελεγκτικό συνέδριο, αλλά πιστεύουμε επίσης, έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι του χρόνου τα πράγματα θα είναι καλύτερα, γιατί ήδη ξεκίνησαν από πέρυσι μεταρρυθμίσεις. Απ' την άλλη όμως, εμείς δίνουμε απαλλαγή για ένα χρόνο σε αυτή την Επιτροπή. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό ποτέ, ότι η απαλλαγή μας αφορά ένα χρόνο, ένα έτος. Οπότε πρέπει να είμαστε σε θέση να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας, να τις παίρνουμε πολύ στα σοβαρά και ανάλογα κάθε έτος να κάνουμε τις προτάσεις μας. Έχοντας όλα αυτά υπόψη, από πλευρά της ομάδας μου, θέλουμε να υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες στην έκθεσή σας. Θα δούμε μήπως μπορούμε να κάνουμε μια διασύνδεση εδώ περισσότερο ορατή από ό,τι είναι τώρα με τις προηγούμενες χρονιές. Επίσης υπάρχουν κάποιοι τομείς όπου η άποψή μας διαφέρει ελαφρά από εκείνη του εισηγητή. Κυρίως το θέμα της έρευνας. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει κάτι θετικό χάρη στη δουλειά που ο Επιτροπός έχει κάνει για να διορθωθεί η κατάσταση όσον αφορά τις δικές του αρμοδιότητες. Τα τελευταία δύο-τρία χρόνια δίνουμε διαφορετικές ε, συστάσεις. Τις έχει ακολουθήσει ο Επίτροπος και μάλιστα έχει πάει και λίγο ακόμα πιο μακριά από ό,τι θα περιμέναμε εμείς, από ό,τι του ζητήσαμε. Ακόμα λοιπόν και αν υπάρχουν προβλήματα ακόμα με την έρευνα, δεν βλέπω ότι θα μπορούσε να έχει κάνει περισσότερο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο διάστημα που μεσολάβησε. Οπότε και εδώ θα έχουμε κάποιες τροπολογίες. Έρχομαι τώρα στο θέμα της απλοποίησης. Πολλά από τα συμπεράσματα που υπάρχουν στην έκθεση είναι ευπρόσδεκτα και θα τα υποστηρίξουμε φυσικά. Όμως είναι αλήθεια επίσης ότι κάποιες από τις πληροφορίες που ζητάτε κύριε Σιγητά υπάρχουν ήδη. Καταλαβαίνω γιατί το ζητάτε, γιατί δεν είναι πάντα εύκολο να τις εντοπίσει κανείς αυτές τις πληροφορίες ή να τις συγκρίνει να τις χρησιμοποιήσει. Όμως ο κύριος Κάλλας έχει δίκιο όταν λέει ότι υπάρχουν. Άρα, μάλλον πρέπει να μιλήσουμε με την Επιτροπή και να συζητήσουμε πώς θα μπορούσαμε να έχουμε ένα καλύτερο σύστημα για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις και να είναι πιο εύκολο για μας να κάνουμε τη δουλειά μας που σημαίνει ότι θα είναι πιο εύκολο και για το κοινό να έχει τις πληροφορίες αυτές εφόσον το επιθυμεί. Υπάρχει και κάτι που θέλω να προσθέσω. Κάτι σχετικά με τη διαφάνεια. Η διαφάνεια για μας πρέπει να είναι ένα από τα κύρια ζητήματα. Και τις προηγούμενες χρονιές το υπογραμμίσαμε. Και στην έκθεση Μιλντερ το λάβαμε υπόψη, βάλαμε ένα ολόκληρο κεφάλαιο. Συμφωνώ βέβαια μαζί σας ότι υπάρχει κάτι σχετικό σε μια παράγραφο εκεί που λέτε ότι πρέπει να έχουμε όλες τις πληροφορίες που θέλουμε Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να προσθέσουμε ότι οι πληροφορίες που έχουμε δεν είναι τόσο καλές ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σύγκριση και ούτε έχουμε και την πλήρη εγγύηση ότι οι πληροφορίες αυτές είναι έγκυρες. Επίσης ότι δεν υπάρχει εγγύηση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβώς τα στοιχεία που έχουμε ζητήσει. Επίσης, θα έπρεπε να συστήσουμε κάτι για την πρόταση για διαφάνεια. Πολλά σχόλια είναι θετικά. Έχουν γίνει βελτιώσεις αλλά μπορούν να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η κατάσταση στο μέλλον. Εξωτερικές υποθέσεις, χρηματοδότηση, εξωτερικές δράσεις. Συμφωνώ με πολλές από τις δηλώσεις των εισηγητών ότι και σε αυτόν τον τομέα είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι το πρώτο βήμα για έναν έλεγχο είναι η πρόσβαση στην ενημέρωση, στις πληροφορίες, στα στοιχεία. Και εδώ δεν είμαστε ακόμα στην καλύτερη δυνατό κατάσταση. Εννοείται ότι θα συνεργαστούμε στενά μαζί σας στη συνέχεια και θα καταφέρουμε να συμφωνήσουμε πάνω σε μια καλή έκθεση την οποία και θα μπορέσουμε να υπερψηφίσουμε και που θα προτείνει την απαλλαγή. Μια τελευταία συμβουλή, αν μου επιτρέπετε. Και εδώ νομίζω ότι θα υποβάλω κάποια τροπολογία γι' αυτό. Ότι η έκθεση να ξεκινάει με τα κύρια συμπεράσματα, τα πιο σημαντικά. Αν διαβάσετε τα έγγραφα που στέλνουμε στο κοινό εμείς, το κοινό δεν υπάρχει περίπτωση να καταφέρει να καταλάβει τίποτα. Αν μη τι άλλο θα πρέπει να διευκολύνουμε τον κόσμο να είναι σε θέση να καταλάβει τι γράφουμε. Ξεκινώντας από τα κύρια συμπεράσματα. Το έχουμε ξανακάνει αυτό στο παρελθόν. Αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε να πετύχουμε και πάλι. Ευχαριστώ. Κυρία Κρέσλε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή διότι πραγματικά τοποθετήθηκε επί της ουσίας. Ε, θέλω να σας πω ότι μετά την αντίδραση του Επιτρόπου ανησυχώ λιγάκι γιατί ε, δεν είμαι σίγουρη κατά πόσον κατάλαβε την ε, καλή μας πρόθεση. Πέρσι είχαμε αυτά που είχαμε και φέτος ε, βέβαια είμαστε πάλι αναγκασμένοι να κάνουμε κάποιες ε, παραχωρήσεις ε, και μάλιστα εκ των προτέρων. Δηλαδή δεν έχει εγκριθεί όλη αυτή η υπόθεση από το Κοινοβούλιο. Γι' αυτό κύριε Επίτροπε θα θέλαμε να ακούσουμε πώς ακριβώς τοποθετήσουμε στα θέματα ουσίας γιατί αυτά τα οποία μας είπατε δεν κατατείνουν στο ότι μας παίρνετε σοβαρά. Παραδείγματο χάρη αυτά που είπατε για τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, το μηχανισμό επαλήθευσης ο οποίος συζητήθηκε και επικρίθηκε για το κατά πόσον είναι αποτελεσματικός ή όχι. Δεν πρόκειται μόνο για τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, πρόκειται και για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τις μελλοντικέ διευρύνσεις. Δηλαδή, δηλαδή πώς θα προετοιμάσουμε στο μέλλον τα κράτη-μέλη να γίνουν, ε, πώς θα προετοιμάσουμε κράτη ώστε να γίνουν κράτη-μέλη της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, το θέμα είναι λοιπόν τι είδου συμπεράσματα εξάγουμε από αυτή τη μεγάλη ήττα και πρόκειται για μια ήττα, ολέθρια ήττα αυτή την οποία υποστήκαμε στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Γι' αυτό λοιπόν ανησυχώ για τον τρόπο, λόγω του τρόπου με τον οποίο αντιδράστε. Θα με ενδιαφέρει επίσης ε, να γνωρίζω ε, το θέμα του name and shame και της ε, κριτικής ε, στα κρατημέλη. Πώς ακριβώς τοποθετήσετε εκεί. Εσείς λέτε έχουμε τις 3.500 σελίδες να τις διαβάσει κανείς την ετήσια δραστηριότητα. Το είπατε και μόνοι σας, είναι 3.500 σελίδες. Εντάξει, εγώ το κοιτάω κατά καιρού, αλλά εμείς θα θέλαμε να έχουμε ένα έγγραφο της Κομισιόν. Γιατί το Annual Activity Report δεν είναι έγγραφο της Κομισιόν, είναι διαχειριστικά έγγραφα. Εμείς όμως θα θέλαμε να έχουμε ένα της Κομισιόν που να ε, απαντά σε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει η έκθεση ε, σύνθεσης ε, αυτή όμως είναι άχρηστη πρέπει να το πω, μια παντελώς άχρηστη έκθεση και εντωμεταξύ το πώς εργάζεται η Κομισιόν αυτό το θεωρώ δεδομένο. Δηλαδή είτε αυτή την έκθεση θα την καταρτίζετε και θα την μετατρέπετε σε ένα πραγματικό έγγραφο το οποίο δίνει πληροφορίες για θέματα διαχείρισης ή θα κάνουμε κάτι καινούριο. Και τώρα αυτό που υπάρχει είναι το να υπάρξει κάτι καινούριο. Ε, παραθέσατε τα διάφορα σημεία, τα έγραψα και εγώ αυτά και δεν είμαι σίγουρη κατά πόσον η δυσφορία του Κοινοβουλίου έγινε κατανοητή σε ορισμένα θέματα. Παραδείγματο χάρη στο θέμα τη πολιτική κτηρίων. Ίσως να μην το πιστεύετε, αλλά αυτά που σα λέω δεν είναι δικά μου, δεν είναι απαραίτητα δικά μου. Δηλαδή, εγώ ε, δεν είμαι η μόνη εκείνη που δουλεύει σε αυτό το εργοτάξιο, λέει χαριτολογώντα η κυρία Κρέσλε. Ω εκ τούτου, ε, θεωρώ ότι πρέπει να ασχοληθείτε με τα θέματα αυτά και εμείς ε, θα προσπαθήσουμε να ε, παρουσιάσουμε τα διάφορα αιτήματα και για κάθε ένα από αυτά τα αιτήματα χρειαζόμαστε μία τοποθέτηση της Κομισιόν. Γιατί αλλιώς εγώ δεν θα μπορέσω να συστήσω στην ομάδα μου να συμφωνήσει. Χρειαζόμαστε μία ε, κατηγορηματική τοποθέτηση της Κομισιόν που θα δείχνει ότι τα παίρνετε όλα αυτά σοβαρά χωρίς να χρειαστεί να καταφύγουμε στα μέσα πίεση στα οποία καταφύγαμε πέρυσι. Η κυρία Λουτσέβα, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, тъй като една голяма част от доклада на, Ένα μεγάλο κομμάτι της εκθέσεως για την απαλλαγή αφορά την Βουλγαρία. Είχαμε δυστυχώ τεχνικό πρόβλημα, υπάρχει φοβερή παρεμβολή στα ακουστικά και είναι αδύνατο να κάνουμε διερμηνία. Δεν ακούγεται ο μιλητή σωστά. Από ό,τι φαίνεται κάποιος εδώ έχει πρόβλημα με την απαλλαγή της Κομισιόν και δημιουργεί παράσιτα και παρεμβολές. Ah. Ξανά αγαπητοί συνάδελφε. Ξανά όμως η παρεμβολή συνεχίζεται. Δυστυχώς δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Έχουμε τεχνικό πρόβλημα.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 Ε, Δυστυχώ δεν, ε, το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει. Είναι ένα φοβερό χαμηλό βόμβο Δεν μπορούμε να ακούσουμε. Λοιπόν, ε, η κυρία θα τα πει στα αγγλικά. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που προσφέρεστε να τα πείτε στα αγγλικά και ελπίζω οι τεχνικοί να λύσουν το πρόβλημα. Αγγλικά μπορείτε? Συμφωνείτε? Λοιπόν, αγγλικά. Ευχαριστώ. Ένα μεγάλο τμήμα της εκθέσεως αφορά την Ουρμανία και τη Βουλγαρία. Γι' αυτό χρειάζεται να πω μερικά πράγματα. Πριν από αυτή την έκθεση επανειλημμένα συζητήσαμε τα προβλήματα της απορρόφησης των ευρωπαϊκών πόρων στην Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Νομίζω ότι οι δημοσιεύσεις σε αυτό τον τομέα δείχνουν ότι η Βουλγαρία πήρε την ετικέτα του κακού, του άτακτου μέλους Ευρωπαϊκής Ενώσεως, του μέλους που δεν είναι σωστό στη συμπεριφορά του. Θα πρέπει η επικοινωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των χωρών αυτών Ρουμανίας και Βουλγαρίας να βελτιωθεί, αλλά όχι με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία μόνο, γιατί αυτό μπορούσε να συμβεί σε όλες τις χώρες και όχι μόνο ε, στις νέες χώρες. Γι' αυτό Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ετοιμάσει κάποια συγκεκριμένα μέτρα προς βελτίωση αυτής της ε, επικοινωνίας. Πέραν αυτού θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιείται η έκθεση σε σχέση με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που πετυχαίνουν οι δύο χώρες αυτές γιατί πολύ Γιατί αν συνεχίσουν στα πράγματα θα εξακολουθεί να θεωρείται η Βουλγαρία ότι δεν είναι σωστή σαν εταίρος. Χρειάζεται πιο συγκεκριμένη διαδικασία. Το λέω αυτό διότι όλοι γνωρίζετε ότι φέτος η Βουλγαρία έλαβε υπόψη όλα τα δέοντα μέτρα για να βελτιώσει την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Στην έκθεση του κυρίου Οντί, για, τον οποίο, για την οποία τον συγχαίρω, βλέπω για πρώτη φορά στην έκθεσή του λοιπόν, όπως έλεγα, συστάσεις απευθυνόμενες προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περί επιμονής και προετοιμασίας των σχέσεων με αυτές τις δύο χώρες, με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Και ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιμείνει επί της βελτιώσεως των αποτελεσμάτων και βελτιώσεως του μηχανισμού εκτελέσεως των προγραμμάτων και ελέγχου αυτών. Υπάρχει αμοιβαία ευθύνη. Αν βασικός υπεύθυνος για την εκτέλεση των προγραμμάτων και απορρόφηση των πόρων είναι η χώρα, δηλαδή η Βουλγαρία. Αυτό ισχύει. Απ' την άλλη όμως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τις δικές της ευθύνες για την όλη διαδικασία. Διότι εγκρίθηκαν πολλές διαδικασίες κατά την προεταξιακή περίοδο όπου η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν στη Βουλγαρία Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι ο νέος μηχανισμός και ένα στρατηγικό έγγραφο για τις χώρες θα είναι κάτι που πρέπει να προετοιμάζεται και για την ένταξη των χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να το προετοιμάζει. Οι χώρες χρειάζονται χρόνο να προετοιμαστούν. Χρειάζονται χρόνο για να δημιουργήσουν δικούς τους μηχανισμούς. Για να μπορέσουν να αντιδράσουν σωστά. Και να απορροφούν και να χρησιμοποιούν σωστά τους πόρους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε λέει Ο κύριος Μούλντο, ο συνάδελφος κύριος Μούλντο έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα προτιμούσα να μιλήσω μετά την Επιτροπή, αλλά εν πάση περιπτώσει, μια που μου δίνετε το λόγο. Πρέπει να μιλήσουμε ακόμα για αυτά, αλλά εγώ δεν μπορώ να είμαι τόσο καθυσχαστικός προς την Επιτροπή όπως ήταν άλλοι. Γιατί πιστεύω ότι υπάρχει προσπάθεια για την αναβολή της απαλλαγής. Και γιατί? Πιστεύουμε ότι η βελτίωση δεν είναι μεγάλη. Γίνεται με αργούς ρυθμούς. Αν δούμε τις βελτιώσεις, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι σε 25 χρόνια θα έχουμε θετική τάση. Προηγουμένως όχι. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και πολύ ενθαρρυντική αυτή η κατάσταση. Δεύτερον, καρδιά της διοργανικής συμφωνίας ήταν ότι θα είχαμε περιλήψεις. Και αν δείτε τι έγινε τα τρία τελευταία χρόνια, τα ψηφίσματα ε, του Κοινοβουλίου τι ζητάνε, θα δείτε τι λένε για τις εθνικές δηλώσεις. Και η Επιτροπή είπε πέρυσι ότι δεν θα το έκανε. Και εμείς τους πιέσαμε και στείλαμε το μήνυμα και τελικά είπαν ότι εντάξει θα το κάνουν. Τελικά όμως, ακόμα και σήμερα, δεν ξέρουμε τι κάνανε. Ακόμα και ο εισηγητής δηλώνει στο σημείο 20 ότι λυπάται για την στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά το ψήφισμα Γιώργενσον το 2008 για την απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2006 όσον αφορά την ποιοτική αξιολόγηση των ετησίων συνόψεων στις εκθέσεις δραστηριότητα. Οπότε, τι περιμένει η Επιτροπή. Να δώσουμε εμεί απαλλαγή. Η ομάδα μου ειλικρινά προβληματίζεται πάρα πολύ. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αγνώρισε πλήρω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το κάνει κάθε χρόνο. Υπόσχεται ότι θα κάνει και τελικά δεν κάνει. Πολύ ωραία λέει ο Πρόεδρος. Ε, νομίζω ότι η Κομισιόν ε, πρέπει να τα λάβει αυτά υπόψη και όποτε θέλει μπορεί να παρεμβεί. Κύριε Μποτόπουλο, έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είχα δύο παρατηρήσεις, κάπως συγκεκριμένες και τεχνικής φύσεως, αλλά θα ήθελα να πω την γνώμη μου σχετικά με αυτά που μόλις ανέφερε ο κύριος Μέλντερ. Καταλαβαίνω την ανησυχία σας, όμως πιστεύω ότι θα ήταν υπερβολή να μην δώσουμε φέτος την απαλλαγή, φέτος που έγινε μια σημαντική προσπάθεια από πλευρά τη Επιτροπής. Το λέει καλά, πιστεύω και ο συγητής, ότι δεν είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι, αλλά ότι έχει γίνει προσπάθεια. Έπειτα, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα εσείς, υπάρχει και ο παράγοντας ευρωπαϊκές εκλογές. Και δεν ξέρω κατά πόσο είναι η καλύτερη χρονιά φέτος να μην δώσουμε απαλλαγή. Εντάξει, έτσι αυθόρμητα αντίδρασα, αντέδρασα σε αυτά που είπε ο κύριος Μέλντερ. Όμως, δύο παρατηρήσεις κάπως τεχνικής φύσεως έχω να κάνω. Επί της ουσίας συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Γιόγκερσεν, που είναι αρμόδιος επί της ουσίας της έκθεσης, που είναι καλή και που με κάποιες μικρές βελτιώσεις μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερη. Ποιες είναι οι παρατηρήσεις μου. Πρώτον, για την Όλαφ. Είναι σημαντικό να μιλήσουμε για την Όλαφ, γιατί αποτελεί μέρος του των μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας για να καταπολεμήσουμε, καταπολεμήσουμε την απάτη. Εγώ διαβάζω άνετα αγγλικά και ελληνικά, αλλά εδώ δεν καταλαβαίνω πολύ καλά. Αν κατηγορείτε την ίδια την όλα όταν λέτε ότι δεν λειτουργεί πολύ καλά ή αν αυτό που θέλετε να πείτε είναι ότι δεν δίνουμε στην αυτά τα μέσα που χρειάζεται για να μπορέσει να δράσει κτλ. Θα ήθελα να, εδώ να γίνετε πιο συγκεκριμένος γιατί η έκθεση Κρέσλερ για την Όλαφ το λέει. Η δεύτερη παρατήρησή μου έχει να κάνει με τις παραγράφους 66, 67 και 68 όπου για πρώτη φορά δεν μιλάμε για το 2007 ενώ η απαλλαγή είναι για το 2007 αλλά μιλάμε για τέτοια 2000-2006 για να κάνουμε έτσι μια πιο σφαιρική ανάλυση για το τι γίνεται με το Ταμείο Συνοχής, το Κοινωνικό Ταμείο κλπ. Δεν είναι τυχαίο που αναφέρεται και η Ελλάδα στο σημείο 67. Εγώ δεν είμαι μεταξύ εκείνων που κάθε φορά που υπάρχει κάποια καταδίκη της χώρας τους αμέσως ε, ξεσηκώνονται. Όχι, αλλά νομίζω ότι εδώ στο 66, 67 και 68, σε αυτά τα τρία σημεία, ε, χρησιμοποιούμε μια διαφορετική μέθοδο. Μιλάμε για μια πιο μακρά περίοδο, έξι ετών, και η Ελλάδα ήταν στις αρχές μόνο τότε του συστήματος. Άλλαξε η κατάσταση από τότε. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν είναι δίκαιο, δεν είναι σωστό να ε, χρησιμοποιούμε εδώ πέρα να μιλάμε για μια συγκεκριμένη χώρα, name and shame όπως λέμε. Είναι άδικο η Κομισιόν ε, θέλει να πει κάτι. Αν δεν θέλει να πει κάτι η Κομισιόν, ο εισηγητής, ο κύριος Οντί, έχει το λόγο για να κλείσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις τους που είχαν την καλοσύνη να μου διαβιβάσουν. Σημείωσα δεόντως το συνέστημα του Αντιπρόεδρου της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής τι απόψει του όσον αφορά την παρέμβαση του συναδέλφου Γιώργενσεν σχετικά με τη βελτίωση κάποιων παραγράφων. Συμφωνώ όσον αφορά τη διαφάνεια, συμφωνώ μαζί σα ότι αυτέ οι παραγράφοι, παράγραφοι θα πρέπει να βελτιωθούν. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ευχαριστώ την κυρία Γκρέσλε και την κυρία Λούτσεβα όσον αφορά τις απόψεις που εξέφρασαν. Όσον αφορά τον συνάδελφο Μόλτερ, είμαι έτοιμος να συνεργαστώ μαζί του αν επιθυμεί κάτι τέτοιο επί κάποιων πτυχών της εκθέσεως νομίζω ότι έχουμε κοινή ανησυχία και εκείνος και εμείς θέλουμε μια θετική δήλωση αξιοπιστίας δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε ότι βελτιώθηκε η κατάσταση το να προτείνει, προτείνουμε τώρα αναβολή της απαλλαγής σημαίνει να μην ψηφίσουμε την απαλλαγή διότι αν Έχουμε κάποια πρόοδο που μερικοί θεωρούν αργή. Η αναβολή για την απαλλαγή γίνεται τον Οκτώβριο. Δεν θα αλλάξει η κατάσταση τον Οκτώβριο συγκρίση με σήμερα. Τον Οκτώβριο θα έχουμε αρνητική ψήφο. Άρα δεν θα διθετήσει τίποτα η αναβολή. Αντιθέτω, θα πρέπει να ζητήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μα πει πώ και πότε θα έχουμε θετική δήλωση αξιοπιστία, γνωρίζοντα βέβαια ότι Ξέταση του κειμένου της συνθήκης ε, μας δείχνει ότι από τη στιγμή που το ελεκτικό συνέδριο, το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζονται το, ε, το ελάχιστο επίπεδο των σφαλμάτων θα μπορέσουμε εμείς σε μια διάσκεψη που προτείνει η έκθεση να θέσουμε επιτάπητος προσυζήτηση τους τρόπους που θα χρησιμοποιήσουμε για να καταλήξουμε σε θετική δήλωση εξοπιστίας και παράγραφος 20 που υπογραμμίζει ο κύριος Μούλτερ για να δικαιολογήσει την αναβολή της απαλλαγής δεν θεωρώ ότι είναι επαρκής βάσης εν συγκρίση με το έβρος των πολιτικών συνεπειών που θα έχει μια τέτοια αναβολή, μια τέτοια απόφαση. Όσον αφορά τα όσα είπε ο συνάδελφος Βοτόπουλος για την Όλαφ είναι η δεύτερη αυτή πτυχή που τονίσατε ότι θέλει η Όλαφ να έχει περισσότερους πόρους και μέσα στη διάθεσή της. Ίσως δεν είναι καλά διατυπωμένο το κείμενο, χρειάζεται κάποια βελτίωση. Όσον αφορά το ότι κατανομάζονται κάποιες χώρες στις παραγράφους περί συνοχής, αν στα πλαίσια συμβαστικής τροπολογίας αντικείμενο συμβασμού διαφόρων μελών ή συμφωνία των σκιωδών εισηγητών αφαιρέσουμε αυτό το στοιχείο που κατανομάζονται οι χώρες, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι χαίρομαι που διεξήχθη αυτή η άκρος επικοδομητική συζήτηση. Σημειώνω τις ανησυχίες κάποιων μελών και επιμένω απευθυνόμαστε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προετοιμασία που θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια είναι επιτακτική ανάγκη κατά την άποψή μου η άκρο ανικανοποιητική αυτή κατάσταση αυτή που συνοψίζουμε επί 9 μήνες στη διαδικασία της απαλλαγής που επί 14 χρόνια οδηγεί σε αρνητική δήλωση αξιοπιστίας και επί 14 χρόνια το Κοινοβούλιο ψηφίζει την απαλλαγή αυτή η κατάσταση λέγω κύριε Επίτροπε πρέπει να συζητηθεί πλήρω στην Ολομέλεια. Θα πρέπει το Κοινοβούλιο να λάβει διαβεβαιώσει ότι κάποια μέρα θα έχουμε θετική δήλωση εξοπιστίας. Κλείνοντα ανεκδοτικά κάπως, εκφράζοντα τι ανησυχίε μου πριν κλείσω τα όσα λέω για την έκθεση. Ένας υπάλληλο μου είπε μία μέρα, φου, τελικά το Κοινοβούλιο γαυγίζει, γαυγίζει δεν δαγκώνει ποτέ. Νομίζω ότι θα πρέπει κανείς να προσέχει, διότι τη στιγμή που το Κοινοβούλιο θα δαγκώσει, θα είναι δύσκολα τα πράγματα για όλους. Δοθέντως ότι πιστεύω ότι είναι και η ώρα όλα να συζητηθούν και ότι θα πρέπει να δοθεί διαβεβαίωση ως εκπρόσωποι των λαών που είμαστε, θα πρέπει να εμφανιστούμε μπροστά μας μπροστά συγγνώμη, στο εκλογικό σώμα και να πούμε ότι ελέγχουμε τον εκτελεστικό κλάδο όσον αφορά την χρήση των πόρων τη ευρωπαϊκή Ενώσεω και εκτελεστική εξουσία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σέβεται την υπόσχεση του Προέδρου Μπαρόζο. Δηλαδή γνωρίζουμε πώς και πότε θα έχουμε τελικά μια θετική δήλωση αξιοπιστίας. Πρόεδρος, ε, σας ευχαριστούμε πολύ και για άλλη μια φορά σας συγχαίρουμε. Δεν έχουμε ολοκληρώσει τις ε, εργασίες. Ε, πρέπει να συνεχιστούν. Ε, πάντως κάνατε πάρα πολύ δουλειά και θα θέλαμε να σας ευχαριστούσουμε για την πολύ καλή δουλειά σας κύριε Οντή. Για να κλείσει λοιπόν αυτό το θέμα, μην ξεχνάτε η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 5η 19 Φεβρουαρίου στις 12 η ώρα. Και δέστε λιγάκι και... Ε, τις ε, άλλες ημερομηνίες. Ε, θα πρέπει λοιπόν την Δευτέρα στις 16 Μαρτίου να ψηφίσουμε εδώ στην Επιτροπή μας. Αν τα πράγματα πάνε άσχημα θα δούμε. Μετά στην Ολομέλεια θα ε, δούμε την έκθεση όντω την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Ωραία. Οπότε περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξη. 6 με 12 μαζί θα τα εξετάσουμε αυτά τα σημεία. Είναι η απαλλαγή για τα άλλα όργανα. Η συγητής είναι ο κύριος Σέντεγκάρτ. Έχετε το λόγο κύριε Σέντεγκάρτ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Στόχος μου και καθήκον μου ήταν να ελέγξω τους λογαριασμούς για τα άλλα θεσμικά όργανα. Δεν είναι και λίγα. Οπότε, αποφασίσαμε να θέσουμε προτεραιότητες. Αποφασίσαμε να εξετάσουμε την απαλλαγή στο Συμβούλιο πρώτα απ' όλα. Και γιατί κάναμε αυτή την επιλογή. Διότι στην Επιτροπή μας πολλές φορές και επανειλημμένως και για χρόνια εκφράζουμε την δυσαρέσκειά μας εξαιτίας της πλήρους αδιαφορίας που δείχνει το Συμβούλιο απέναντι στο δικό μας το έργο, τη δικιά μας τη δουλειά. Που είναι να ελέγχουμε την χρήση των πιστώσεων και των κονδυλίων και να βλέπουμε κατά πόσο η χρήση τους γίνεται με υπεύθυνο τρόπο ή όχι. Πριν από μισή ώρα είχαμε ένα παράδειγμα, ένα ξεκάθαρο παράδειγμα έχουμε εκπροσώπους του Συμβουλίου εδώ και πριν φτάσουμε στους λογαριασμούς του Συμβουλίου, τι κάνουν, φεύγουν από την αίθουσα. Να λοιπόν, τελικά, πώς γίνεται ο διάλογος ανάμεσα σε εμά και το Συμβούλιο. Αυτό το σημερινό γεγονός αποτελεί κατάφορη απόδειξη της έλλειψης διαλόγου που έχουμε με το Συμβούλιο. Αντί να είναι εδώ, και να μπορούμε να συζητήσουμε και να κρίνουμε κατά πόσο οι απαντήσει του είναι ικανοποιητικέ, αν πρέπει να υπογραμμίσουμε το ένα ή το άλλο, αν είναι εντάξει λογαριασμοί. Δεν φτάνουμε σε αυτό. Για το Συμβούλιο δεν υπάρχει τίποτα. Δεν έρχεται καν να συζητήσει μαζί μα. Πόσο μάλλον να απαντήσει. Η συζήτηση θα ήταν ε, εκτός κατηγορίας αν μιλούσαμε εδώ πέρα για αθλητικά γεγονότα. Οπότε πού θα οδηγήσει η σημερινή συζήτηση που κάνουμε εδώ μεταξύ μας, τη στιγμή που δεν υπάρχει διάλογος με το Συμβούλιο. Είναι απόν. Αυτό το οποίο εγώ επιθυμώ είναι πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις συζητητές από τις διάφορες ομάδες, να ευχαριστήσω τη γραμματεία επίσης γιατί η συνεργασία μας ήταν πάρα πολύ καλή. Και επίσης να αναφερθώ λιγάκι στο ιστορικό, να κάνω μια ιστορική αναδρομή. Ορισμένοι πιστεύουν ότι η έκθεση αυτή είναι αρκετά αδύναμη, ότι υπάρχει δυνατότητα απόρριψης της απαλλαγής και μπορεί κανείς να αναρωτηθεί τελικά η έκθεση αυτή είναι αρκετά έντονη, δεν είναι αρκετά έντονη. Ακούγονται όλα. Ε, λοιπόν, η έκθεση αυτή αποτελεί τη συνέχεια, επιμένω σε αυτό, τη συνέχεια της στάσης που η Επιτροπή μας έχει οθετήσει τα τελευταία χρόνια. Το 2002, εδώ δηλαδή και καιρό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από πρόταση της δικιάς μας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής πρότεινε ψήφισμα για την απαλλαγή 2000 για το Συμβούλιο. Και, συνεχίζει στα αγγλικά όμιλη της, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο κατά το παρελθόν δεν ήλεγξαν την εφαρμογή των διαφόρων τμήματων του προπολογισμού. Το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι βάσει της ε, της αυξανόμενης χρήσης κονδυλίων από το διοικητικό προπολογισμό του Συμβουλίου και στις εξωτερικές δράσεις και την ασφάλεια και την άμυνα, τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις, στόχος του διακανονισμού πρέπει να αποσαφανιστεί έτσι ώστε να υπάρχει διάκριση ανάμεσα στις παραδοσιακές και διοικητικές δαπάνες όλους αυτούς τους νέους τομείς πολιτικής συνεχίζει στα δανέζικα ο μιλητής. Συνεπώς οι θέσεις αυτές έχουν επανεληφθεί από το Κοινοβούλιο και ξανά και το 2007 μετά από πρόταση της δικιάς μας Επιτροπής στη διαδικασία απαλλαγής για το Συμβούλιο και το 2005 όπου το Κοινοβούλιο και πάλι στα αγγλικά ο μιλητής για μεγαλύτερη διαφάνεια στον τομέα της κοινή εξωτερικής πολιτικής ζητάει από το Συμβούλιο σύμφωνα με το σημείο 42 στην Διοργανική Συμφωνία να φροντίσει ώστε δεν υπάρχουν δαπάνες από την κατηγορία αυτή στον προϋπολογισμό και επιφυλάσσεται να αναλάβει τα σωστά διαβήματα εφόσον η συμφωνία αυτή παραβιαστεί. Συνεπώς, πέρυσι στην έκθεσή μας ε, γράψαμε για την απαλλαγή 2006 ότι το Συμβούλιο δεν υπέβαλε ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων στο Κοινοβούλιο και ζητάμε από το Συμβούλιο να ξαναδεί την απόφαση του αυτή, να την αναθεωρήσει και να μας στείλει έκθεση δραστηριοτήτων ώστε να διαπιστωθεί ότι λογοδοτεί όντως για ε, τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Ήταν πάντα ξεκάθαρο λοιπόν τα τελευταία χρόνια η Επιτροπή μας, το Κοινοβούλιο ολόκληρο, έχουμε επιμείνει ξανά και ξανά. Θέλουμε εμείς ως εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών να παίρνουμε την αποστολή μας πολύ στα σοβαρά και να φροντίζουμε τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογούμενων να δαπανώνται σύμφωνα με τις αποφάσεις που έχουν υιοθετηθεί. Αυτό είναι κάτι που ισχύει και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φυσικά το ίδιο και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και για το Συμβούλιο εννοείται. Δυστυχώς όμως διαπιστώνουμε ότι το Συμβούλιο εμένει στη θέση του, εμένει στη στάση του να μην θέλει να συζητήσει με τη δικιά μας Επιτροπή. Προφανώς και θέλουμε να εγκρίνουμε τους λογαριασμούς και να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες ε, σφάλματος, αλλά θα πρέπει να είμαστε σε θέση να εξετάζουμε τις διάφορες θέσεις. Υπάρχει ένα παράδειγμα που αναφέρεται, είναι τα ταξιδιωτικά έξοδα. Πρόκειται για την 2022 ε, γραμμή που αναφέρεται στα έξοδα διερμηνίας. Εδώ οι 66% μεταφέρθηκαν από ε, την διερμηνία στα ταξιδιωτικά έξοδα στον τομέα της ε, εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. 66% το 2006 το ποσό αυτό ξεπερνούσε τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Πάνω από 12 εκατομμύρια ευρώ μεταφέρθηκαν από την θέση διερμηνία στη θέση ταξίδια. Γιατί? Γιατί δεν μπορούν να βρεθούν χρήματα αλλού. Γιατί είναι ένα μυστήριο όλα αυτά τα ταξίδια. Τόσο σημαντικό ποσό. Να μην μπορούμε να το εξετάσουμε. Ίσως να υπάρχει μια πολύ καλή εξήγηση. Αλλά μας χρειάζεται αυτή η εξήγηση και αυτή την εξήγηση δεν μπορούμε να την πάρουμε γιατί το Συμβούλιο δεν επιθυμεί να μας τη δώσει, δεν επιθυμεί να συζητήσει για αυτό το θέμα. Ανταυτού διαπιστώνουμε ότι το Συμβούλιο δεν αποκρίνεται στην πρόσκλησή μας να έρθει και να συζητήσει με τους σκιώδες εισηγητές και με μένα τον ίδιο τον εισηγητή. Αντίθετα το Συμβούλιο αρνείται να δώσει έκθεση όσον αφορά την εκτέλεση των πιστώσεων και ούτε έχει δώσει πλήρη έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο. Εγώ τουλάχιστον ως εισηγητής έτσι το βρίσκω. Και συμφωνώ με τον Πρόεδρό μας, ο οποίος είπε ότι ο έλεγχος του προπολογισμού είναι ένα βασικό στοιχείο για την αξιοπιστία ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει δηλαδή πάρα πολύ μεγάλη σημασία πώς χρησιμοποιούμε τα χρήματα του φορολογούμενου. Αν δεν υπάρχει λοιπόν έλεγχος προπολογισμού που να αξίζει το όνομά του, οι πολίτες δεν θα εμπιστεύονται τα ευρωπαϊκά κοινοτικά όργανα. Συνεπώς πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας τώρα που είμαστε τις παραμονές των ευρωεκλογών. Είναι δύσκολο να λέμε ότι είμαστε εντάξει. Δεν είναι δυνατόν να μας πιάνουν όμοιρους με αυτόν τον τρόπο, να μας ζητάνε να εγκρίνουμε τους λογαριασμούς χωρίς να παίρνουμε τις απαντήσεις που θέλουμε. Δεν λέω ότι πρέπει να απορρίψουμε την απαλλαγή αναγκαστικά. Όχι, εγώ αυτό που θέλω είναι μια κατάσταση που να μας οδηγήσει στο να εγκρίνουμε τους λογαριασμούς, αλλά να έχουμε τις πληροφορίες που ζητάμε. Θα μπορούσαμε λοιπόν για μια τελευταία φορά, αυτή είναι η πρότασή μου, να προσπαθήσουμε, έχουμε ήδη προσπαθήσει τρεις-τέσσερις φορές, ένα ξανά προσπαθήσουμε και πέμπτη φορά, ώστε αυτά τα θέματα που παραμένουν σε κρεμότητα για μας να τα ζητήσουμε από το Συμβούλιο, να έρθει το Συμβούλιο και να μας δώσει απαντήσεις. Κατά πόσο θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα δεν ξέρω, αλλά τουλάχιστον κανείς δεν θα μπορεί να πει ότι δεν κάναμε μια προσπάθεια παραπάνω. Από εκεί και πέρα, τα απαντήσετε όχι το Συμβούλιο, θα πρέπει να πάρουμε κάποια απόφαση για την τελική ψηφοφορία που θα έχουμε το Μάρτιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σιγητά. επεξεργαζόμαστε το Συμβούλιο, έχουμε και τους άλλους. Για την ώρα συζητούμε το Συμβούλιο, έχουμε πολλά να πούμε για το Συμβούλιο προφανώς. Ίσως θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από το Συμβούλιο να μας πει κάτι σε αυτή τη φάση. Το Συμβούλιο πριν το ελεγκτικό συνέδριο. Ας ακούσουμε. Ο κ. Συγητής κάτι θέλει να πει. Ορίστε. Πρόεδρε, έχω... Μετά θα ασχοληθούμε με τα άλλα. Πρώτα το Συμβούλιο, μετά τους υπόλοιπους. Δεν υπάρχει πρόβλημα, λέει ο πρόεδρος. Ορίστε. Λοιπόν, το Συμβούλιο έχει κάτι να πει. Όχι. Ωραία. Το συνηθίσαμε αυτό. Τι έκανα. Απλώς ε, επιβεβαιώνει αυτό, αυτό που λέει ο εισηγητής. Δεν μπορούμε να κρύψουμε τίποτα. Δεν μπορούμε να κρύβουμε χρήματα από τους φορολογούμενους μας. Τα κράτη-μέλη μπορούν. Τι γίνεται με το ελεκτικό συνέδριο, έχουν τίποτα να πούν οι εκπρόσωποι του ελεκτικού συνεδρίου, τα κράτη-μέλη. Καλώς. Ο κύριος Βοτόπουλος και ο κύριος Πόμεζουρή. Ο κύριος Βοτόπουλος πρώτος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ω κοιόδη εισηγητή τη ομάδα των Σοσιαλιστών πάνω σε αυτό το σημαντικό το θέμα, αυτή τη σημαντικότατη έκθεση, Πρέπει να πω απευθυνόμαστε στον ειδηγητή ότι η σοσιαλιστική ομάδα συμφωνεί απόλυτα με την τοποθέτησή του και θα ήθελα επίσης να προσθέσω δύο λόγους για τους οποίους θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό επιτέλους να μας δώσει κάτι το Συμβούλιο. Να πω επίσης το ότι απουσιάζει το Συμβούλιο τώρα ε, δικαιώνει όλους μας που επί σειρά ετών λέγουμε ότι κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει να αλλάξει το όλο θεσμικό πλαίσιο, κυρίως σε θέματα όπως είναι η ασφάλεια και η άμυνα. Να μιλάμε μια φωνή το Συμβούλιο και να μην κρύβεται κάθε φορά πίσω από την εναλλασσόμενη Προεδρία και να λέει ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσει η επόμενη Προεδρία. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Προτρέχω. Λοιπόν, θα ήθελα να αναφέρω άλλους δύο λόγους τα όσα είπε ήδη ο εισηγητής που υποστηρίζουν ότι πρέπει τώρα να πάρουμε απάντηση από το Συμβούλιο. Λοιπόν, για ποιο λόγο, πρώτα απ' όλα, η περίφημη αυτή η συμφωνία κυρίων που αναφέρθηκε επανειλημμένα και κανεί, οι περισσότεροι μάλλον δεν την έχουμε δει, ε, δημιουργεί κι άλλο ένα πρόβλημα. Κανεί δεν φαίνεται να το αναφέρει. Δηλαδή, αν είχε υπογραφεί τη δεκαετία του 70, τη δεκαετία του 70 δεν είχαμε καμία δαπάνη όσον αφορά την ασφάλεια και την άμυνα είναι ένας νέος ε, τομέας ο οποίος θα πρέπει να καλυφθεί. Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από συμφωνία κυρίων της δεκαετίας του 70 ενώ αναφερόμαστε σε νέα πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Πέραν αυτού, θα έλεγα ότι τώρα οι τρέχουσες εξελίξεις με τις συνθήκες της Αβώνας που ελπίζουν ότι κάποτε και σύντομα καλύτερα να τεθεί σε ισχύ get αλλάξει πλήρως το θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά την ασφάλεια και τις εξωτερικές σχέσεις. Αν δεν κάνουμε τώρα την αλλαγή, αν δεν πάρουμε τώρα απαντήσεις, νομίζω ότι αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρό κίνδυνο να χάσουμε τελείως όταν ο νέος ύπατος εκπρόσωπος θα αρχίσει θα πάρει τη θέση του με νέο γραφείο με νέες υπηρεσίες και τα επόμενα λίγα έτη δεν θα γνωρίζουμε ακριβώς ποιος είναι υπεύθυνο γιατί. στα θέματα ασφαλείας και αμήνης. Είναι πολύ σημαντικό τώρα να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά. Σωστά τα είπε ο εισηγητής. Είναι ενδιαφέροντα και σημαντικά αυτά που είπε. Δεν θέλουμε να συμμετάσχουμε στη διαμόρφωση πολιτικής, ζητούμε να γνωρίζουμε για ποιο λόγο, παραδείγματο χάρη, έχουμε μεγαλύτερες ταξιδιωτικές δαπάνες και αυτό είναι κάτι που αφορά τη δουλειά μας, τη δουλειά των βουλευτών. Αφορά το θεσμικό μας έργο. Και αν δεν πάρουμε απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Είναι τόσο απλό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λέει ο κύριος Θα εξετάσω από, τον κύριο, από αυτό που είπε και ο κύριος Σοντή Πού είναι το Συμβούλιο? Συμβούλιο. Τίποτα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν εκεί οι ταμπέλες που λένε Council. Είναι εδώ απλώ για να παρακολουθούν τη συζήτηση για την έκθεση οντί και να μεταφέρουν αλλού το τι λέμε εδώ. Και όμως το Συμβούλιο είναι ένα πολύ σημαντικό θεσμικό όργανο και για τον ε, έλεγχο προπολογισμού επίσης είναι πολύ σημαντικό θεσμικό όργανο. Όχι, το κινητό μου φταίει. Καλά, να το απομακρύνω γιατί ακούγεται κάποιο ήχο στο μικρόφωνο. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικό θεσμικό όργανο. Πού το λοιπόν. Ο Επίτροπο Κάλλα, που σίγουρα έχει ένα σωρό υποχρεώσει, και όμω ήρθε και κάθισε στη συζήτηση που έγινε για την έκθεση οντί. Τώρα είσαι από το Συμβούλιο. Συμβούλιο φάντασμα. Εγώ θα ήθελα, αν μη τι άλλο, να περάσει στο Συμβούλιο το ότι η στάση αυτή του Συμβουλίου απέναντι στο Κοινοβούλιο εαμάν πια. Δεν μπορούμε να δεχτούμε πια μια τέτοια στάση. Εμείς είμαστε η αρχή του προπολογισμού ε, λοιπόν, το Συμβούλιο πρέπει να έρχεται εδώ και να λογοδοτεί. Δεν μπορεί να έχει αυτή τη στάση που έχει. Είναι θλιβερό. Να είναι απόν ή να είναι παρόν αλλά να σιωπά. Γιατί το αποτέλεσμα είναι ότι δεν απαντάει στις ερωτήσεις του εισηγητή. Πρέπει να έχουμε μαζί συναντήσεις εργασίας Χρειάζεται συνεργασία μεταξύ μας δηλαδή για να δούμε θα εγκρίνουμε ή δεν θα εγκρίνουμε τους λογαριασμούς του Συμβουλίου. Ε, λοιπόν, εμείς κάνουμε ένα σωρό προσπάθειες για να έχουμε διάλογο μαζί τους. Και διάλογο έχουμε με όλα τα υπόλοιπα όργανα, στα οποία θα δώσουμε ή δεν θα δώσουμε απαλλαγή, από το πιο μικρό ευρωπαϊκό οργανισμό μέχρι την Επιτροπή. Όλοι μας ανοίγουν τα γραφεία τους, όλοι είναι σε επαφή μαζί μας, τηλεφωνικά ή αλλιώς, όλοι εκτός από το Συμβούλιο. Πολύ σωστά λέγατε ότι η συμφωνία κυρίων του 70 για μένα με ξενίζει κάπως, διότι το Κοινοβούλιο πρέπει να ζητάει το κείμενο επειδή αυτό αναφέρεται μόνο σε μία πράξη του Συμβουλίου. Όταν υπάρχει τέτοια συμφωνία κυρίων αφορά δύο πλευρές. Για να ισχύει πρέπει να είναι γνωστή αυτή η συμφωνία εκατέρωθεν. Αν είναι κάτι που έχει συντάξει μία πλευρά μόνο και μόνο εκείνη γνωρίζει και εμείς δεν ξέρουμε τίποτα, ε, τότε τι να το κάνουμε, να μας λείπει. Στο κάτω-κάτω μπορεί να λέει το Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να απαντάει στο Κοινοβούλιο. Ξέρω εγώ τι λέει. Πού το. Πού είναι. Σε ποια πράξη του Κοινοβουλίου αναφέρεται αυτό ή τελικά είναι ένας μύθος που εμείς πρέπει να δεχτούμε και ό,τι λέει το Συμβούλιο πρέπει να το δεχόμαστε. Ε, όχι, αν υπάρχει τέτοια συμφωνία, ε, πούντι να μας λένε ότι υπάρχει τέτοια συμφωνία, αλλά είναι κάπου που εσείς δεν μπορείτε να τη βρείτε, ε, για όνομα. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να αμφισβητήσει κανείς τα πάντα. Λοιπόν, εδώ καταγγέλλω επίσημα αυτήν την υποτιθέμενη συμφωνία των υποτιθέμενων κυρίων. Γιατί πούντι. Στηρίζω λοιπόν, όπως και ο σοσιαλιστής συνάδελφος, τον εισηγητή στη διαμαρτυρία του αυτή. Που επαναλαμβάνουμε. Γιατί ξανά και ξανά, μετά τη Λισαβόνα, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει επίσης ώρες να συζητάνε. Και αν μη άλλο το Συμβούλιο πρέπει να συμπεριφέρεται υπεύθυνα απέναντι στους πολίτες. Συνεπώς, ελπίζω, οικετεύω, ζητάω από το Συμβούλιο να ανταποκριθεί στις εκκλήσεις μας τις τόσο σημαντικές, για τόσο σημαντικά θέματα. Γιατί δεν είναι δυνατόν, όσο σημαντικό και αν είναι το Συμβούλιο, να περνάει και να ξεφεύγει από τον έλεγχο της αρχής του προπολογισμού. Δεν γίνεται. Πρέπει να έρθει και να απαντήσει. Συνεπώς, ο εισηγητής έχει τη δικιά μου την προσωπική στήριξη, την πολιτική στήριξη και ζητάω για άλλη μια φορά να μην κρύβεται το Συμβούλιο πίσω από τέτοια άλοθη τέτοιων υποτιθέμενων συμφωνιών, αλλά να αναλάβει τις ευθύνες του και να έρθει να απαντήσει στις ερωτήσεις του εισηγητή και της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ. Ah, Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Οντί έχει το λόγο, παρακαλώ. Είναι μια κατάσταση πολύ δύσκολη και ενοχλητική. Από τις φήμες που άκουσα στους διαδρόμους, κατάλαβα ότι αυτή η συμφωνία κυρίων αφορούσε τον προϋπολογισμό. Δηλαδή όσον αφορά τις προβλέψεις δαπανών υπήρχε ένας αμοιβαίος σεβασμός των θεσμικών οργάνων, αλλά όχι όσον αφορά την εκτέλεση. Εδώ πρόκειται περί εκτελέσεως του προϋπολογισμού που συζητούμε. Άρα η συμφωνία κυρίων δεν αφορά την εκτέλεση, αυτή θα πρέπει να υποβάλλεται στη διαφάνεια, στην επιταγή για διαφάνεια εναντί των πολιτών. Και μήπω, διερωτώ με Πρόεδρε, μήπω θα πρέπει στην Ολομέλεια να υποβληθεί προφορικό ερώτημα στο Συμβούλιο. Συμβολικό πώ. Για να πούμε ότι θέλουμε να εξηγηθεί επί του θέματο. Διότι καταλαβαίνω τι θέση του συγγητού εγώ. Αν χρησιμοποιήσουμε τη διαδικασία απαλλαγή για να διευθετήσουμε το θέμα να ξεκαθαριστεί μεταξύ Συμβουλίου και μόνο δεν ξέρω αν είναι κάτι σωστό. Τελευταίο. κάτι διαδικαστικό. Δεν κατάλαβα ποια είναι η άποψη του συγητή. Βλέποντας το κείμενο που έχουμε στους φακέλους υπάρχουν εκρεμή σημεία. Προτείνει αναβολή ο εισηγητής. Τι θα υποβληθεί σε ψηφοφορία. Ο καθένα θα υποβάλει τροπολογία και στο τέλο θα κάνουμε συμβαστικέ τροπολογίε. Τι θα γίνει διαδικαστικά, αυτό ρωτάω. Διαδικασία που ακολουθήσουμε, ποια θα είναι. Κύριε Κάμρη, ευχαριστώ. μα τελειώνει ο χρόνος. Χάνουμε την υπομονή μας με αυτή την στάση του Συμβουλίου. Μήπως υπάρχει κάποια λύση, εσείς σαν πρόεδρος της Επιτροπής μας, να πείτε στο Συμβούλιο, κοιτάξτε, αν δεν έρθετε να συζητήσουμε, θα πρέπει να αρνηθούμε τη χορήγηση απαλλαγής. Δεν μπορούμε να επομιστούμε ευθύνε αν δεν συζητήσουν μαζί μα και αν δεν απαντήσουν ερωτήσει μα. Ουσιαστικά έναν κίνδυνο διατρέχουν να μην τους δώσουμε απαλλαγή. Υποθέτω ότι θα ερχόταν εάν τους κάνατε αυτή τη δήλωση εσείς. Äh, Πρόεδρος, ε, Αύριο λοιπόν ε, θα συζητήσουμε για το θέμα αυτό στις πολιτικές μας ομάδες και νομίζω ε, η Επιτροπή εδώ ε, συμφωνεί, συμφωνούν όλοι, δηλαδή δεν μπορούμε να εμφανιστούμε στους φορολογούμενους και όλα αυτά τα εκατομμύρια τα οποία δαπανώνται για νέες πολιτικές να μην ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Νομίζω αυτό δεν είναι δυνατόν να λάβει η χώρα. Ε, γιατί αν το κάνουμε αυτό τότε να μοιράζουμε και επιταγές. Ε, λευκές επιταγές. Κύριε Σιγητά, έχετε το λόγο για να κλείσουμε παρακαλώ αυτό το θέμα. Και νομίζω ε, ετέθηκε ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα του συναδέλφου κυρίου Οντή σχετικά με τις τελίτσες ναι, θα ήθελα να απαντήσω στον κύριο Οντί να απαντήσω στο συγκεκριμένο ερώτημα που έθεσε. Αυτό που θέλουμε είναι να υποβάλουμε δύο τροπολογίες. Μία τροπολογία στην οποία χορηγούμε την απαλλαγή και μία άλλη τροπολογία στην οποία την αρνούμεθα. Και πιστεύω και νομίζω ότι υπάρχει υποστήριξη γι' αυτό, ότι για μία ακόμη φορά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ζητήσουμε από το Συμβούλιο να απαντήσει, να απαντήσει στις ερωτήσεις μας. Και όταν θα διεξαχθεί η ψηφοφορία τον Μάρτιο, νομίζω ότι για πολλούς αυτό που θα έχει αποφασιστική σημασία θα ήταν αν θα έχει απαντήσει στα ερωτήματά μας το Συμβούλιο ή δεν θα έχει απαντήσει. Οπότε έχουμε τις δύο δυνατότητες. Μέχρι το Μάρτιο και μπορούμε να δώσουμε πέμπτη ή έκτη ευκαιρία στο Συμβούλιο να απαντήσει στις ερωτήσεις μας και να συμπεριφερθεί σωστά. Όσον αφορά τη Συμφωνία Κυρίων, θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να απευθυνθείτε στις διάφορες κυβερνήσεις σας ο καθένας από εσά για να μάθουμε αν υπάρχει αυτή η Συμφωνία Κυρίων. Διότι αν υπάρχει μια τέτοια συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τότε όλες οι κυβερνήσεις των κρατών μελών θα πρέπει να είναι ενήμερες. Δεν είναι το Συμβούλιο που θα ήξερε κάτι διαφορετικό. Διότι εκεί είναι εκπρόσωποι των κρατών μελών. Άρα θα πρέπει ο καθένας από εμά στο κοινοβούλιο του ή στην κυβέρνησή του να το ξεκαθαρίσει να δει κατά πόσο γνωρίζουν οι κυβερνήσει ότι υπάρχει αυτή η συμφωνία κυρίων. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κατάλληλα για την υποστήριξή σα. Νομίζω ότι συμφωνούμε εν γέννη αν ε, η Επιτροπή μα πρέπει να διαδραματίσει ένα ρόλο σαν εκπρόσωπο των πολιτών όσον αφορά τον έλεγχο του προπολογισμού και πώ χρησιμοποιούνται τα χρήματα των φορολογουμένων θα πρέπει να έχουμε τι αναγκαίε πληροφορίε Διαφορετικά δεν έχει νόημα αυτή η δουλειά. Πρόεδρος, ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, πράγματι θα δώσουμε χρόνο στο Συμβουλίο μέχρι την επόμενη συνεδρίαση. Προτείνω δηλαδή τη 10η Μαρτίου. Μέχρι τότε ε, θα πρέπει να έχουν καταθέσει προτάσεις τους. Και κύριε Ισηγητά, αυτή η υποτιθέμενη συμφωνία κυρίων, κοιτάξτε, είναι τόσο παλιά που ρίχνοντας έτσι εδώ μια ματιά μόνο οι συνάδελφοι Κρέσλε, Μούλντα και ο μόνο αυτοί την ε, γνωρίζουν. Γιατί όλοι οι άλλοι, ε, τα κράτη τους δεν ήταν καν ε, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε τώρα για την εποχή της ΕΟΚ. Έξι κράτη που ήταν ιδρυτικά κράτη της ΕΟΚ. Πάμε στο επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης. Κύριε Ισηγητά. Ευχαριστώ πολύ. Το επόμενο σημείο αφορά το δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Προτείνουμε να δώσουμε την απαλλαγή στο Γενικό Γραμματεία του, Γραμματέα συγγνώμη, του Δικαστηρίου για την περίοδο 2007. Υπάρχουν κάποιες θετικές εξελίξεις όσον αφορά τα λογιστικά. Θα ήθελα να πω κάποια πράγματα. Για πρώτη φορά δημοσίευσε το δικαστήριο τις διοικητικές δαπάνες για το 2007 και δεύτερον, ακόμα και αν υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την διαρμηνία και τους ειδικού για την πληροφορική υπάρχει μια σχετική αναφορά στο ειδικό προσωπικό. Υπάρχει θετική εξέλιξη άλλη ότι μειώθηκε η διάρκεια της διαδικασίας παρόλο που παραμένει κάποιο ανησυχητικό στοιχείο. Δηλαδή υπάρχει μια αύξηση τις υποθέσεις του πρωτοδικείου και μετά στην έκθεση δραστηριοτήτων το δικαστήριο συμπεριλαμβάνει ένα κεφάλαιο που παρουσιάζει το ποια συνέχεια δόθηκε σε πρώτερες αποφάσεις του Κοινοβουλίου περί απαλλαγής. Ε, όλα αυτά είναι πάρα πολύ θετικά και θα συστήσουμε και στα άλλα θεσμικά όργανα να το κάνουν και θα αναφερθώ και στις άλλες περιπτώσεις αργότερα. Θα ήθελα να συγχαρώ λοιπόν το δικαστήριο γι' αυτό και θα ήθελα να επιμείνω ούτως ώστε αυτή η δήλωση προϋπολογισμού που δόθηκε από τα μέλη του δικαστηρίου όσον αφορά τα οικονομικά του συμφέροντα να δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δικαστηρίου. Θα πρέπει να διοριστεί και ένας ανεξάρτητος ελεγκτής που θα πρέπει να συντάσει έκθεση όσον αφορά τις δηλώσεις που παρελήφθησαν. Είναι σημαντικό στοιχείο που θα εξασφαλίζει μια παρακολούθηση και αξιόπιστο έλεγχο. Είμαστε θετικοί και ελπίζω και το δικαστήριο να είναι θετικό όσον αφορά την, ε, τις επιθυμίες που θα εκφράσουμε σχετικά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ε, ας προχωρήσουμε. Νομίζω ε, καλύτερα να τα πάρουμε όλα μαζί. Ε, τα αποτελέσματα που είχαμε μέχρι τώρα ήταν ιδιαίτερα θετικά. Ε, κύριε Σιγητά, πάμε στο 8, στο ελεγκτικό συνέδριο. Μάλιστα. Είναι το επόμενο σημείο, το ελεκτικό συνέδριο και εδώ προτείνουμε να χορηγηθεί η απαλλαγή, να δοθεί στο Γενικό Γραμματέα του Ελεκτικού Συνεδρίου για το έτος 2007. Βεβαίως ε, με την ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι υπάρχει έκθεση αξιολογήσεως που συνετάχθη το Δεκέμβριο του 2007 που δείχνει ότι το σύστημα διαχειρίσεως των διοικητικών δαπανών ταιριάζει με τις διεθνείς προδιαγραφές. Ταυτόχρονα ελπίζουμε αυτές οι διεθνείς λογιστικές προδιαγραφές να πετύχουν τελικά το στόχο τους. Σημειώνουμε με ικανοποίηση ότι τα μέλη του ελεκτικού συνεδρίου δίνουν μια δήλωση όσον αφορά τα οικονομικά του συμφέροντα και τα περιουσιακά του στοιχεία, αλλά λυπούμεθα διότι αυτές οι δηλώσεις είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα. Και επαναλαμβάνουμε την ευχή μας αυτές οι δηλώσεις να είναι προσβάσιμες, να είναι σε ένα δημόσιο μητρό που θα ε, βρίσκεται στο διαδίκτυο και προτείνουμε και το διορισμό ενός ανεξαρτήτου ελεγκτού επιφορτισμένου να αναφέρει και να προβάλλει κάθε χρόνο τις δηλώσεις που υποβάλλονται. Και τέλος, το ελεκτικό συνέδριο στον στην έκθεση δραστηριοτήτων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει ένα κεφάλαιο όπως ζητήσαμε και από το δικαστήριο, κάτι που έκανε, ένα κεφάλαιο που λεπτομερώς θα δείχνει α, τι συνέχεια δόθηκε στις αποφάσεις περί απαλλαγής που έδωσε τα προηγούμενα χρόνια το Κοινοβούλιο και ελπίζουμε να το δεχτούν αυτό στο Ελεκτικό Συνέδριο, σημείο 9, Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή και εκεί προτείνουμε να χορηγηθεί η απαλλαγή. Η έκθεση εμπεριέχει σειρά θετικών παρατηρήσεων σχετικά με την επιτευθύσα πρόοδο κατά την περίοδο που πέρασε, αλλά έχουμε και κάποιες συστάσεις. Παραδείγματος χάρη, σημειώνουμε ότι τα μέλη της ΟΚΕ δεν δημοσιεύουν τις δηλώσεις τους οικονομικών συμφερόντων ή πληροφορίες σχετικά με άλλες δραστηριότητές τους, μισθωτές ή μη μισθωτές δραστηριότητες. Και γι' αυτό ε, συστήνουμε όλα τα μέλη να υπέχουν την υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση όσον αφορά τα συμφέροντά τους και προτείνουμε και το διορισμό ανεξαρτήτου ελεγκτού. Άλλο σημείο, η έκθεση δραστηριοτήτων είναι πολύ ποιοτική των ετησίων δραστηριοτήτων. Στην επόμενη έκθεση θα θέλαμε να μας εξηγούν όμως ε, πώς η Οικονομική, και Οικονομική Επιτροπή αντέδρασε βάσει των προτέρων συστάσεων του Κοινοβουλίου. Είτε έκανε κάτι, αν είναι κάτι θετικό, είτε δεν έκανε το παραμικρό. Αλλά να μας εξηγήσουν γιατί δεν έκαναν κάτι και θα πρέπει να το ξανασυζητήσουμε αυτό. Και ελπίζουμε ότι και εκεί η αντίδραση είναι θετική όσον αφορά την Επιτροπή των Περιφερειών. Θα επανέλθουμε αργότερα διότι υπάρχουν πράγματα να πούμε. Είμαστε στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή στο σημείο 11 και εκεί προτείνουμε την χορήγηση της απαλλαγής ε, για το έτος 2007 αναφέρουμε σειρά θετικών εξελίξεων παραδείγματο χάρη ο διαμεσολαβητής της 14 Δεκεμβρίου Α, να το βρω, να το βρω. Συγγνώμη, λέει ο αγορητής. Ο διαμεσολαβητής της 14 Δεκεμβρίου του 2007 υιοθέτησε μία απόφαση σχετικά με την ετήσια δήλωση του διαμεσολαβητή όσον αφορά τα συμφέροντα, τα οικονομικά συμφέροντα, τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων. Και αυτή δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα αυτή η δήλωση, στην ιστοσελίδα του διαμεσολαβητή. Θεωρούμε ότι είναι θετικό επίσης ότι στις 2 Ιουνίου του 2008 ο διαμεσολαβητής προσεχώρησε στη Διοργανική Συμφωνία της 25ης Μαΐου του 1999 που είχε συνηφθεί μεταξύ Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις εσωτερικές έρευνες που πραγματοποιούνται από την Όλαφ. Όσον αφορά το διαμεσολαβητή ζητούμε επίσης στην επόμενη έκθεση δραστηριοτήτων του να συμπεριλαμβάνεται ένα κεφάλαιο που θα παραθέτει λεπτομέρειες σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στις αποφάσεις απαλλαγής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα προηγούμενα ετή. Και τέλος, και φτάνω στο σημείο 12 τώρα, ο Ευρωπαίος Ελεκτής για την προστασία των δεδομένων και εδώ προτείνουμε και σε αυτό το φορέα να δοθεί η απαλλαγή και εκεί έχουμε θετικέ ε, εξελίξει όσον αφορά τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασία Δεδομένων. Υποστηρίζουμε θετικέ εξελίξει, αλλά για μία ακόμη φορά, όπω και σε άλλου προηγούμενους τομείς. Ζητούμε στην επόμενη έκθεση δραστηριοτήτων του φορέα αυτού να συμπεριλαμβάνεται ένα κεφάλαιο που θα αναφέρεται λεπτομερώς στη συνέχεια που δόθηκε στις αποφάσεις περί απαλλαγής προηγουμένων ετών που, δόθηκαν, που ελήφθησαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρακτικά θα πρέπει η δουλειά που κάνουμε κάθε χρόνο να είναι μια δουλειά συνεχής να υπάρχει συνέχεια, να μπορούμε να προδεύουμε χάρη στις διασυνδέσεις που υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων εκθέσεων. Ελπίζω επίσης ότι η απάντηση θα είναι θετική και από την πλευρά του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας των Δεδομένων. Αυτά και ευχαριστώ. Äh, Κύριε Σιγητά, το 10 τώρα να το εξετάσουμε ξεχωριστά ή να το πάρουμε μαζί την Επιτροπή των Περιφερειών. Ναι, αλλά μπορούμε ε, να τα πάρουμε όλα μαζί. Ορίστε. Συνεχίζει ο συγητής. Η Επιτροπή των Περιφερειών, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να εξεταστεί ξεχωριστά. Εγώ τουλάχιστον έτσι εκλαμβάνω την όλη κατάσταση. Ε, Πάμε στους ε, οργανισμούς εξαιρουμένης της Επιτροπής των Περιφερειών. Θέλει κάτι να πει το ελεγκτικό συνέδριο ή οι οργανισμοί ελέγξαν πάρα πολλά θετικά. Βεβαίως ε, και εσείς ε, βρίσκεστε εδώ για να ρωτηθείτε. Πάντως ο εισηγητής ε, νομίζω ότι στο σχέδιο της εκθεσής του ήταν ιδιαίτερα φιλικός απέναντι σε εσά. Άρα δεν θέλει κανείς ε, να λάβει το λόγο. Κλείνει αυτό το θέμα. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε εισηγητά και πάμε τώρα στο σημείο υπαριθμών 10. Η... Τι θέλετε να κάνουμε με το 10? Κυκλισμένων των θυρών, τότε καλύτερα ε, να προτάξουμε τα άλλα θέματα και αυτό να τα αφήσουμε στο τέλος. Εντάξει, πολύ ωραία τότε έκλεισε αυτό το σημείο της ημερησίας διάταξης και θα ήθελα να επανάλαβω για τους ε, συναδέλφους την 5η 19 Φεβρουαρίου στις 12 η ώρα όπως και για όλες τις άλλες εκθέσεις είναι καταλεκτική ημερομηνία για την υποβολή των τροπολογιών. Πάμε τώρα στα σημεία 13 και 14 και μετά στο 10 και κλεισμένων των θυρών. Ε, σημείο υπαριθμών 13 παρακαλώ. Ειδική έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου ε, αριθμός 9 ε, 2008 σας το διαβάζω στα αγγλικά όπως το αναφέρει το Κοκομπή σχετικά με την αποτελεσματικότητα της υποστήριξης Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης για την Λευκορωσία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία. Ε, η συγγήτρια είναι η κυρία Λούπτσεβα και εκ μέρους του ελεγκτικού συνεδρίου έχουμε τον κύριο Ουσκέβιτς. Ε, κύριε Ουσκέβιτς, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, Mitglied des Rechnungshofes und einen wichtigen Tagesordnungspunkt. Herr Uskewitsch, bitte. Thank you. Thank you very Λοιπόν, ευχαριστώ, λέει ο κ. Σοσκίεβιτς. Ευχαριστώ που μου δίνετε δυνατότητα να σας παρουσιάσω την ειδική έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της υποστήριξης Ευρωπαϊκής Ενώσεως τομείς της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης για τη Λευκορωσία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία. Το ελεκτικό συνέδριο ανέλαβε αυτή, αυτό τον έλεγχο λόγω της μεγάλης σημασίας του ζητήματος και τη σχετικότητα του ελέγχου όσον αφορά το, να βοηθήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμόσει τη νέα πολιτική γειτονία και το σχετικό μέσο. Μετά τη διεύρυνση που έγινε το 2004 και το 2007, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε νέου γείτονε, τη Μολδαβία, την Ουκρανία και τη Λευκορωσία, μεταξύ άλλων. Και σε αυτέ τι σημαντικέ μεθοριακέ χώρε, με πάνω από 60 εκατομμύρια κατοίκου, θέματα ελευθερία, ασφαλεία και δικαιοσύνη καταπολέμηση της ε, ελεύκανσης χρήματος, ε, παρανόμου ε, διακίνησης ατόμων κλπ. Είναι διάφορα θέματα που πρέπει να εξεταστούν προς όφελος αυτών των χωρών και προς όφελος των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Η πολιτική αστάθεια και η διαφθορά ε, έκαναν, δημιούργησαν προβλήματα, δυσκόλεψαν αυτή την πολιτική και έγινε και κατεπίγουση ανάγκη επιβολής της πολιτικής. Μεταξύ του 2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάλαβε τη σημασία που έχει αυτή η περιοχή και γι' αυτό διέθεσε 166 εκατομμύρια ευρώ για τη Λευκορωσία, για συγκεκριμένους τομείς. Έλεγχο των συνόρων και διαχείριση αυτών, μετανάστευση, διαχείριση του ασύλου, καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και τέλος ε, δικαστικούς τομέας και ορθή διακυβέρνηση. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, το ελεκτικό συνέδριο εξέτασε το πρόγραμμα που κόστιζε περίπου 100, ε, 100 ε, εκατομμύρια ευρώ. Τα 100 από τα 166 που σας είπα. Και ήθελα να απαντηθούν και τα εξή ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα ήταν σε ποιο βαθμό η ευρωπαϊκή υποστήριξη για τα προγράμματα για ασφάλεια, δικαιοσύνη ε, ήταν επιτυχή στη Λευκορωσία. Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι για ενδεχόμενη ε, ε, υποεφαρμογή των προγραμμάτων. Σε ποιο βαθμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαδικασία εκμάθησης για να λαμβάνει υπόψη τα μαθήματα για τη συνέχεια της βοήθειας στον τομέα της ελευθερίας, της ασφαλείας και της δικαιοσύνης. Βλέποντας τους στόχους του ελέγχου μπορούμε να κάνουμε τις κάτωθοι παρατηρήσεις που έγιναν και οι παρατηρήσεις αυτές. Λοιπόν πρώτα απ' όλα ένα μεγάλο κομμάτι των ελέγχων πέτυχε ικανοποιητικά αποτελέσματα, όμως ήταν περιορισμένο το πεδίο εν συγκρίση με την κλίμακα των προβλημάτων που θα αντιμετωπιστούν. Καμιά φορά μπορούμε να πούμε ότι ήταν σταγόνα στον ωκεανό εν συγκρίση με τις πραγματικές ανάγκες. Η καλύτερη απόδοση ήταν στον τομέα της διαχειρίσεως των συνόρων. Η υποστήριξη υποστήριξε τη βελτίωση του ελέγχου και τη δημιουργία δυναμικού για τον έλεγχο των συνόρων στι χώρε. Ιδιαίτερα επιτυχή ήταν η βοήθεια στη Μολδαβία και την Ουκρανία, εξαιρετική αποστολή. Δυστυχώ, οι, οι επιδόσεις ήταν μία ικανοποιητικέ όσον αφορά το άσυλο και τη μετανάστευση. Η πρόοδο για το χορήγηση καταφυγίου στου ετούντε άσυλο και του μετανάστε σύμφωνα με τι διεθνεί προδιαγραφέ για ανθρωπιστική αντιμετώπιση ήταν ιδιαίτερα αργή ρυθμή στην Ουκρανία το βλέπουμε στο πλαίσιο 5 του πίνακα. Ε, για τη μετανάστευση, για τη χύση των μεταναστών, για την Ουκρανία. Δείχνουμε εκεί τα αποτελέσματα. Συνέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί με 3,8 εκατομμύρια ευρώ. Και τι θέλαμε να κάνουμε. Να δώσουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό σε εγκατάσταση θετιωτικές για να γίνεται υποδοχή μεταναστών για περίπου 1.600 άτομα το Νοέμβριο του 2006, όταν έγινε ο έλεγχος, τίποτα δεν είχε γίνει. Και ο αριθμός των θέσεων που είχε σχεδιαστεί αρχικά είχε μειωθεί κατά χίλιε από τον αρχικό αριθμό που είχαν προβλέψει για τη στέγαση των μεταναστών. Η Ουκρανία έχει συμφωνία επανεισδοχή με την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει σύντομα να στεγάσει εκατοντάδες και χιλιάδες παράνομους μετανάστες. Τα άλλα αποτελέσματα, ανάμεικτα αποτελέσματα πετύχαμε όσον αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος καθώς και όσον αφορά την, το δικαστικό τομέα και την ορθή διακυβέρνηση. Καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Σε συνεργασία με τα τελωνία, τους μεθοριακούς φύλακες, μυστικές υπηρεσίες, και ήταν ανεπαρκής αυτή η συνεργασία και ανεπαρκής η δίωξη. Και γι' αυτό δεν πήγαμε καλά στον τομέα. Και η σωστή διακυβέρνηση επηρεάστηκε από μακροσκελείς διακασίες δικαστικές και ε, διοικητικές. Και επίσης το είδαμε και στο πρόγραμμα για την καταπολέμηση του ξεπλήματος χρήματος. Με αυτό το πρόγραμμα δημιουργήσαμε μονάδα στη χώρα για να εξετάζεται οικονομικά. Είναι όμως η αρχή. Και είναι προϋπόθεση για την καταπολέμηση του ξεπλήματος χρήματος, η δημιουργία της μονάδας. Για να πετύχουμε καλά αποτελέσματα η σωστή δίωξη και η σωστή νομοθεσία. Βασικός λόγος για τη μην καλή επίδοση στον τομέα αυτό ήταν η έλλειψη σωστής προσπάθειας της χρηματοδότησης από τις εθνικές αρχές. Και έτσι υπονομεύτηκε η βιωσιμότητα του προγράμματος. Να υπογραμμίσω αυτή την παρατήρηση. Να σας δείξω το λέω αυτό. συνεχώς αντιμετωπίζαμε αυτό το πρόβλημα στους ε, ελέγχους όταν βλέπαμε τι γίνεται με την υποστήριξη που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις γειτονικές χώρες. Το καλύτερο παράδειγμα η σύσταση στην έκθεση τι λέει. Λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υποστηρίξει τα προγράμματα όπου το πραγματικό συμφέρον της χώρας αποδέκτου είναι σαφές και είναι εθνικό συμφέρον. Και πρέπει να είναι αλληλεστικό ο στόχο που τίθεται. Και θα πρέπει να είναι και σωστή περίοδο εφαρμογή των προγραμμάτων. Το θέμα είναι η βιωσιμότητα των τελικών αποτελεσμάτων που τυχαίνει το πρόγραμμα, αφού λήξει επίσημα τυπικά η εφαρμογή του προγράμματος. Ποια αποτελέσματα μένουν. Δεύτερο λόγο για τη μην καλή επίδοση. Ε, ε, ε, οι διεθνεί οργανισμοί δεν εφαρμόζουν σωστά τα προγράμματα διότι υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά τις προμήθειες, μακροσκελής διαδικασίες κλπ. και καθυστερούν τα προγράμματα. Και τα συμβαλόμενα μέρη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερμηνεύουν διαφορετικά το διοικητικό και το οικονομικό πλαίσιο από την αιγίδα του ΟΗΕ. Και έτσι εμποδίστηκαν και οι έγκαιρε συνάψει των συμβάσεων και σωστή έλεγχη. Οι χώρε αποδέκτε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν συντόνισαν σωστά την υποστήριξη που δόθηκε από πολλού άλλου δωρητέ και αυτό πολύ συχνά το συναντάμε. Και το παρατηρεί το ελεκτικό συνέδριο. Η συνύπαρξη πολλών οικονομικών μέσων για τον ίδιο σκοπό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και η έλλειψη συντονισμού μεταξύ αυτών παρεμπόδισε τα προγράμματα. Ανεπαρκές εργατικό δυναμικό της αντιπροσωπείας στο Κίεβο που εφαρμόζει τα προγράμματα και τα ελέγχει τα προγράμματα και κυρίως στη Μολδαβία και στη Λευκορωσία. Τέλος, το ελεγκτικό συνέδριο παραδέχτηκε ότι εξωτερικοί παράγοντες υπήρξαν. Πολιτική αστάθεια, πίν. Και αυτοί οι εξωτερικοί ε, παράγοντες επίσης μείωσαν τα αποτελέσματα των ε, προγραμμάτων που εκτελέστηκαν. Ένα καλό παράδειγμα κακής επιδόσεως των προγραμμάτων λόγω πολιτικής αστάθειας και ανεπαρκούς συντονισμού των δωρητών ήταν το πρόγραμμα χρηματοδότησης Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της διαφθοράς. Αυτά τα προγράμματα τα σχετικά είχαν σαν στόχο τη βοήθεια θέσπιση νομοθεσ... στη θέσπιση νομοθεσίας. Το Υπουργείο δικαιοσύνη δεν το ήθελε αυτό όμως, διότι άλλαζε συχνά η κυβέρνηση στην Ουκρανία. Και ενεπλέκονται και άλλοι δωρητέ στον τομέα. Η τη νομοθεσία δεν ανταποκρίνονται στι προδιαγραφέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Λοιπόν, τα μαθήματα που πήραμε είδαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εκμεταλλεύτηκε πλήρω τι δυνατότητες που υπήρχαν να ανταποκρίνονται στα νέα προγράμματα οι των παλιών για να μην επαναλαμβανόνται τα σφάλματα. Να πω μερικά λόγια για τις συστάσεις μας, τις βασικές μας. Ξεχωριστές συστάσεις έχουμε για κάθε ερώτημα ελεγκτικό κάθε θέμα ελεγκτικό. Ένα παράδειγμα σας δώσω. Μία σύσταση από κάθε μία από τις τρεις ομάδες συστάσεων. Πριν να δοθούν και άλλοι πόροι για κέντρα για τους μετανάστες τους παράνομους και για τους ετούντες άσυλο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είναι σίγουρη ότι η κυβέρνηση αποδέκτης θα πληρώσει πράγματι για το τρέχον κόστος, το κόστος λειτουργίας των κέντρων αυτών, ούτω ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα των κέντρων αυτών μετά τη λήξη των προγραμμάτων. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αυξήσει το προσωπικό της στον τομέα της ελευθερίας δικαιοσύνης και ασφάλειας στη Μολδαβία και τη Λευκορωσία και την Ουκρανία και να υπάρχει επαρκής τεχνογνωσία όσον αφορά την προμήθεια και τα έργα που απαιτούνται στι προμήθειε. Και τέλο, όταν ετοιμάζονται νέα προγράμματα, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη συστηματικά, συστηματικότερα μάλλον, ε, παλαιών προγραμμάτων. Στον τομέα, το κεφάλαιο των μαθημάτων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη περισσότερο στην ετοιμασία, προετοιμασία κάποιων κειμένων. Θα πρέπει να υπάρχουν προδιαγραφέ στη χορήγηση δωρεών, κοινέ προδιαγραφέ για τι δωρεέ από διεθνεί φορεί να πω επίση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι αντίθετη όσον αφορά τις, ε, τα πορίσματά μα και τι συστάσει μα. Κάποιε από τι συστάσει μα ήδη έχουν εφαρμοστεί και οι περισσότερε από αυτέ ελπίζουμε ότι θα χρησιμοποιηθούν εν τη εφαρμογή του μέσου για την ευρωπαϊκή, για την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία εταιρική έσω, όχι μόνο για τη Μολδαβία και την Ουκρανία και τη Λευκορωσία, αλλά και για τι άλλε χώρε που καλύπτουν αυτό το μέσο. Να πω επίσης ότι αυτός ο έλεγχος είναι απλώς ε, ένας από τους ελέγχους του ελεκτικού συνεδρίου που έχει σαν στόχο να βοηθήσει την εφαρμογή των προγραμμάτων της ευρωπαϊκής πολιτικής και της πολιτικής γειτονίας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Κάποια προβλήματα που είχαν αναγραφεί παλαιότερα από το ελεκτικό συνέδριο αντικατοπτρίζονται και σε αυτό τον έλεγχο. Να συνοψίσω ότι οι δικαιούχες αρχές ε, δεν είναι τόσο θερμές όσον αφορά την εφαρμογή και την υποστήριξη των προγραμμάτων. Δεν υπάρχει σωστό συντονισμό των δωρητών, υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την ερμηνεία των οικονομικών συμφωνιών μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ηνωμένων Εθνών και τέλος κάτι εξίσου σημαντικό, πολύ συχνά δεν είναι πολύ ορατά τα προγράμματα αυτά της Ευρωπαϊκής Ενώσεω. Τέλος, να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το προσωπικό τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίω εκείνου της αντιπροσωπείας του Κιέβου, που συμμετείχαν στον έλεγχο. Τους ευχαριστώ για την έξοχη ε, συνεργασία και τη βοήθειά του. Ευχαριστώ. Äh, Κοιτάξτε, θα ήθελα να δώσω το λόγο σε ευθύ αμέσω στην εισηγήτρια την κυρία Λούτσεβα Μήπω ε, μήπως μπορείτε να μιλήσετε αγγλικά γιατί υπάρχει πρόβλημα με τα βουλγαρικά. Αν όμω μπορείτε να μιλήσετε αγγλικά μπορούμε να συνεχίσουμε. Παρακαλώ κυρία συνάδελφα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο για την έκθεση αυτή. Γιατί πραγματικά είναι μια πολύ εύστοχη έκθεση. Και θα ήθελα να πω ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα καλή έκθεση η οποία λαμβάνει υπόψη της όλα ε, τα αποτελέσματα που προέκυψαν ε, στις ε, χώρες που μας ενδιαφέρουν. Οι χώρες αυτές, η Ουκρανία, η Μολδαβία και η Λευκορωσία είναι χώρες που έχουν σύνορα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμένα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα έκθεση για τον εξής λόγο. Έχω ε, αποκομίσει εμπειρία στη δική μου τη χώρα πριν από την ένταξη και είχα λοιπόν την ευκαιρία να συγκρίνω τα προβλήματα που είχαν σωρευθεί στη δική μου τη χώρα με τα προβλήματα ε, σε αυτές τις τρεις χώρες κατά τη διάρκεια ε, εφαρμογής ε, των κοινοτικών προγραμμάτων. Ε, Πρόκειψαν λοιπόν ε, διαφορετικά αποτελέσματα σε κάθε μία από αυτές τις τρεις χώρες. Μερικά από αυτά είναι ικανοποιητικά, αλλά πάλι όχι. Και το βασικότερο που μπορεί κανείς να ισχυριστεί ως διαπίστωση είναι ότι οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, οδήγησαν εν γέννη σε θετικά αποτελέσματα. Θα έλεγα λοιπόν ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχουμε και άλλες ε, προτάσεις πέρα από αυτές του ελεγκτικού συνεδρίου έτσι ώστε να βελτιωθεί η χρήση των κοινοτικών κονδυλίων σε ε, χώρες που επιθυμούν να ενταχθούν πλήρως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα λοιπόν να υπάρξει μία σε βάθος ανάλυση των αιτίων που οδήγησαν σε αδυναμίες και ελλείψεις σε ορισμένα προγράμματα γιατί αυτό ε, θα βοηθήσει ε, στην εφαρμογή των ε, προγραμμάτων στο μέλλον. Συστήνω και προτείνω να υπάρχει καλύτερος έλεγχος των, ε, της ε, χρήσης των κοινωτικών κονδυλίων και νομίζω ότι η Κομισιόν πρέπει να είναι πιο ευέλικτη στη χρηματοδότηση προγραμμάτων ε, με κοινοτικά κονδύλια, να χρησιμοποιεί κριτήρια, συγκρίσιμα κριτήρια, έτσι ώστε να λαμβάνεται υπόψη η οικονομική και κοινωνική κατάσταση σε κάθε μία από τις χώρες αυτές. Εξάλλου, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζοντας με απόλυτη σαφήνεια τις υποχρεώσεις της χώρας αποδέκτης μετά το πέρας της εκτέλεσης του κοινωτικού προγράμματος. Σημασία λοιπόν έχει να ε, γίνεται αποτελεσματικότερος έλεγχος ε, των διαφόρων ε, οικονομικών μέσων, να υπάρχει αυστηρότερος έλεγχος από τους διεθνείς οργανισμούς. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε σωστό συντονισμό με εθνικές ΜΚΟ και διεθνείς οργανισμούς ε, οι εθνικές ΜΚΟ να αποκομίσουν ε, θετική εμπειρία και να μπορούν να εφαρμόσουν τις ε, βέλτιστες πρακτικές. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό να συστήσουμε στην Κομισιόν να βελτιώσει την επικοινωνία της με τις κυβερνήσεις των τριών αυτών χωρών. Εξάλλου είναι πολύ σημαντικό να εκταμιευθούν κονδύλια στις χώρες αυτές για διοικητικές δαπάνες. Εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικό ορισμένες από αυτές τις προτάσεις να συμπεριληφθούν στην έκθεση απαλλαγής γιατί εκείνο που παίζει ρόλο είναι να μάθει κανείς από την εμπειρία άλλων κρατών. Μαθαίνει κανείς από ε, χώρες που αντιμετώπισαν προβλήματα κατά την προενταξιακή περίοδο. Αυτό είναι σημαντικό για υποψήφιες χώρες και μόνο αυτό, αλλά εξοικονομούνται και κοινωνικά κονδύλια και οποτεδήποτε αυτά εκταμιεύονται, εφαρμόζονται, ε, χρησιμοποιούνται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μήπως ο κύριος Γκρέι, η Κομισιόν, επιθυμεί να λάβει το λόγο. Θα ήθελα μόνο να υπογραμμίσω, λέει ο Πρόεδρος, ότι αν δείτε λιγάκι την έκθεση ΟΝΤΗ, θα ε, δείτε ότι η ειδική έκθεση του 2009 ήδη περιλαμβάνει τις ε, προτάσεις αυτές της εισηγήτριας και του κυρίου Οντί. Ε, νομίζω ότι είναι τα σημεία 117 έως 138. Είμαι ο Μάρκος Κονάου, είμαι ο αρμόδιος διευθυντής για την πολιτική καλής γειτονίας. Εκ μέρους της ε, Κομισιόν να σας πω ότι εμείς ε, χαιρετίζουμε την έκθεση αυτή κατατίθεται στη σωστή χρονική στιγμή, ε, χρησιμεύσε πάρα πολύ στο να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων και βλέπουμε ότι τα περισσότερα από τα σχόλιά μας ελήφθησαν υπόψη. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ ε, που συμφωνούμε όλοι στο ότι πρόκειται για ένα κανθόδες θέμα. Ε, βεβαίως εδώ ε, μπαίνουμε στην καρδιά της εθνικής κυριαρχίας και παρεμβαίνουμε σε μια δύσκολη, σε μια λεπτή πολιτική στιγμή της ε, Ουκρανίας αλλά και των άλλων ε, κρατών. Ας μην ξεχνάμε ότι εμείς είχαμε την παρέμβασή μας όταν η επίσκεψη της αντιπροσωπείας μας στη Μολδαβία δεν είχε ακόμα ολοκληρωθεί. Η διαχείριση των συνόρων είναι το καλύτερο από ό,τι βλέπουμε στην έκθεση και η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, η δικαιοσύνη, η ε, χρηστή διακυβέρνηση. Αυτά είναι που το μίσο που έχει σημειωθεί πρόοδος. Πρόοδος εξάλλου υπάρχει και στο θέμα της ε, χορήγησης ε, ασύλου. Έχω τη χαρά λοιπόν να σας αναφέρω ότι από τότε που καταρτίστηκε η έκθεση και μέχρι σήμερα μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε, να εξαλείψουμε αρκετές αδυναμίες. Ε, βεβαίως ε, χαιρόμεθα και για τον τρόπο με τον οποίο διατυπώνονται οι συστάσεις, κυρίως όσον αφορά ε, στο ότι πράγματι είναι απαραίτητο να ενταθεί ο διάλογος έτσι ώστε να καταστεί ορατή η μεταρρύθμιση αλλά και να βελτιωθούν οι δυνατότητες. Αυτή είναι η τομή όπου πιστεύουμε ότι από τότε που καταρτίστηκε η έκθεση πράγματι κατορθώσαμε να ε, σημειώσουμε καλύτερα αποτελέσματα. Με μεγάλη μου χαρά άκουσα το ότι θα πρέπει να κάνουμε καλύτερη χρήση της εμπειρίας ε, ε, των, που συνέλεξαν κράτη κατά την προενταξιακή περίοδο πράγματι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την εμπειρία των 12 κρατών μελών. Αυτό θα μας βοηθήσει για να αποκτήσουμε αξιοπιστία είμαι στη διάθεσή σας ε, για περιττέρα σχόλια, αλλά σε γενικές γραμμές κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το λόγο. Εμείς είμαστε ικανοποιημένοι με την ουσία αυτής της έκθεσης και όλα τα άλλα στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι συμφωνούμε οι περισσότεροι επ' αυτού. Ευχαριστούμε το ελεγκτικό συνέδριο, ε, την εισηγήτριά μας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Νομίζω ότι εδώ τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Από ό,τι βλέπω και κανένα μέλος δεν θέλει να λάβει το λόγο. Πάμε στο ε, πρώτο τελευταίο σημείο. Έχουμε μέχρι τις 6,5 χρόνο, το ξέρετε, πρόκειται για την ειδική έκθεση 8 2008 του Ελεγκτικού Συνεδρίου που φέρει την επικεφαλίδα «Είναι αποτελεσματική η πολιτική της ε, πολλαπλής συμμόρφωσης». Ο εισηγητής μας έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η έκθεση που σας παρουσιάζω σήμερα εξετάζει την εφαρμογή της πολιτικής της πολλαπλής συμμόρφωσης, όπως τη λέμε. Είναι πολύ σημαντικό να διαπιστώσουμε εδώ ότι με την εισαγωγή του συστήματος των ενιαίων πληρωμών και με την αποσύνδεση της ενίσχυσης από την παραγωγή, η πολλαπλή συμμόρφωση, δηλαδή οι προϋποθέσεις για την χρηματοδότηση, είναι και η μόνη δικαιολογία για τις ενισχύσεις. Πληρώνονται λοιπόν οι εκμεταλλεύσεις προκειμένου να συντηρούν αυτά τα δημόσια αγαθά που είναι το περιβάλλον και η δημόσια υγεία, όπω επίση και η ευημερία των ζώων. Η πολλαπλή συμμόρφωση λοιπόν αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο τη νέα κοινή γεωργική πολιτική που έχει να κάνει με 50 εκατομμύρια ανθρώπου και 40 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο. Οι παρατηρήσει του ελεκτικού συνεδρίου λοιπόν δεν έχουν να κάνουν τόσο με την αρχή τη πολιτική αυτή, αλλά με την εφαρμογή τη. Και μια που περνάει και η ώρα θα προσπαθήσω κάπως γρήγορα να συνοψίσω την έκθεση αυτή. Πάντως νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να επιμείνουμε σε ένα βασικό στοιχείο, ότι δηλαδή το ελεγκτικό συνέδριο σήμερα θεωρεί ότι έχει γίνει σημαντική πρόοδος, αλλά ότι μένει να γίνει ακόμα μεγάλη πρόοδος, τόσο από την Κομισιόν όσο και από τα κράτη-μέλη, ώστε η πολιτική αυτή πολλαπλής συμμόρφωσης να έχει και αποτελέσματα. Οι υποχρεώσεις που έχουν οι παραγωγοί για να έχουν τις ενισχύσεις δεν είναι κάτι το αρκετά